Commissioner Designate, may I congratulate you on your Να σας συγχαρώ για τη θαυμάσια ομιλία σας όσον αφορά το χρόνο και μακάρι και τα μέλη του Κοινοβουλίου να ακολουθήσουν το παράδειγμα σας. Ο Αντρέας Φόμπ από το ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε Άνσιπ, κύριε υποψήφιε επίτροπε, που είσαστε και Πρωθυπουργό της Εστονίας. Στη χώρα σας επί εννέα έτη ως Πρωθυπουργός μια ολόκληρη σειρά ηλεκτρονικών πρωτοβουλειών αναλάβατε που οδήγησε σε περισσότερες συναλλαγές ηλεκτρονικά και σε μεγαλύτερη εφαρμογή ηλεκτρονικά στη διοίκηση των εφαρμογών αυτών. Η πρώτη μου ερώτηση αφορά ότι τώρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το οποίο θα επιβεβαιωθείτε σε σχέση με τους ε, πρώην συναδέλφου σα, θα βρεθείτε απέναντί του, Μιλήσατε για την κυβερνοασφάλεια. Ήμουν ο ίδιος εισηγητή και μπορώ να σας πω την προηγούμενη εβδομάδα σε μια επίσημη συνάντηση των Υπουργών. Κανένας ε, υπουργό δεν ήταν πρόθυμος να ταξιδέψει προς αυτή τη συνάντηση και γι' αυτό η εντολή για την κυβερνοασφάλεια θα είναι απόλυτα αναγκαία και θα πρέπει να γίνει. Λείπει λοιπόν αυτό το οποίο εσείς αναφέρατε από την Εσθονία να είναι πεισμένοι οι άνθρωποι και οι πολίτες. Τι θα κάνετε ώστε η ενιαία εσωτερική αγορά να μπορέσει να ενισχυθεί σε σχέση με αυτή τη συνιστόσα. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε περιγράφοντας την κατάσταση στην Εσθονία. Θα ήθελα όμως να πω ότι δεν μπορεί η Εστονία, δεν είναι τέλεια ώστε να δώσει μαθήματα σε άλλους. Ένα πράγμα είναι λοιπόν η εφαρμογή κάποιων ψηφιακών θεμάτων στην Εστονία και ένα τελείως διαφορετικό πράγμα είναι τι θα γίνει και τι μπορεί να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφιακά. Η κυβερνοασφάλεια είναι ένα θέμα προστασίας και άμυνας και όπως περιέγραψα στην εισαγωγική μου παρέμβαση οι πολίτες μας υφίστανται πλήγματα από κυβερνοεπιθέσεις λόγω του ότι αυτές οι κυβερνοεπιθέσεις ε, είναι, έχουν το χαρακτήρα του κυβερνοεγκλήματος σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη υπάρχουν οι φορείς για την κυβερνοασφάλεια. Σε κάποια όμως κράτη-μέλη ακόμα δεν υπάρχουν οι φορείς αυτοί για να καλύψουν τα θέματα κυβερνοασφάλειας. Και το ίδιο σε σχέση με τις διάφορες ε, εταιρείες. Ακόμα και μεγάλες εταιρείες δεν έχουν τη δική τους ε, κυβερνοασφάλεια από πλευράς υπηρεσίας. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προετοιμάσει ήδη μια οδηγία και πιστεύω ότι αυτό είναι τεράστια σημασίας, έχει τεράστια σπουδαιότητα. Να αποκτήσει σάρκα και οστά, να γίνει πραγματικότητα η Εστονία υπέστη κυβερνοεπιθέσεις ε, από το, το 2007 και από το 2007 έκτοτε γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι αυτή η άτυπη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ε, υπευθύνων και ε, ηλεκτρονικών εγκεφάλων. Πολλές επιθέσεις τότε είχαν τεράστιες επιπτώσεις και λοιπόν είναι τεράστια σπουδαιότητα να μπορέσουμε να δράσουμε. Ευχαριστώ. Από την, ε, τους σοσιαλδημοκράτες έχετε τον λόγο εσείς παρακαλώ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, θα ήθελα να επικεντρωθείτε το τι συνεπάγεται για την ψηφιακή οικονομία, για τις επιχειρήσεις και το βιομηχανικό τομέα αυτή η συνιστόσα. Μπορεί να υπάρξει ένα νέο δυναμικό, αλλά θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι σημαντικές επιπτώσεις στις εταιρείε ε, και για τις ε, θέσεις απασχόλησης. Χρειάζεται μια νέα πολιτική επενδύσεων και δράσης ε, Ερώτησή μου, πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτές τις επιπτώσεις σας στην αναδιάρθρωση βιομηχανιών και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε αυτή τη φάση για την προς την ψηφιακή οικονομία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω στην πρόοδο στεναρά. Και η πρόοδος πάντα δημιουργεί περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Δεν καταστρέφει θέσεις απασχόλησης, αλλά δημιουργεί περισσότερες θέσεις απασχόλησης η ψηφιακή, το ψηφιακό θεματολόγιο μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις απασχόλησης από ό,τι μπορεί να απολεστούν ή να καταστραφούν. Τα ψηφιακά βρίσκονται παντού. Δεν είναι σωστό να κάνει, λόγο, να κάνει λόγο κανείς σήμερα για τον ψηφιακό τομέα, γιατί όλες οι οικονομίες μας έχουν ψηφιοποιηθεί απόλυτα σήμερα ήδη. Και τα ψηφιακά υποστηρίζουν και την επαναβιομηχανοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως βλέπουμε, ο κύκλος ζωής των προϊόντων ε, έχει συντμηθεί, είναι συντομότερος και κατά τη διάρκεια 2002-2006 υπήρχαν δημοφιλείς τάσεις ε, σχετικά, αλλά τώρα κάνουμε λόγο για την ε, ανάπτυξη την ψηφιακή και τα ψηφιακά σίγουρα θα υποστηρίξουν την αναδιάρθρωση αυτή και μέρος της ε, δημιουργικότητας ε, και της ε, δημιουργίας όσον αφορά τα προϊόντα μας έχουμε πολύ μεγαλύτερο δυναμικό σήμερα από ότι πριν από 10 χρόνια μέσω αυτών των δράσεων. Και πιστεύω λοιπόν ότι η ψηφιοποίηση σίγουρα τελεσίδικα θα υποστηρίξει την επαναβιομηχανοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τούτων λεχθέντων τα ψηφιακά τα ίδια θα προσθέσουν 4% ετήσια στην ανάπτυξη, όταν θα μπορέσουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε την αυθεντική ενιαία εσωτερική αγορά ψηφιοποιημένη. Και έτσι όλοι μπορούμε να υποφεληθούμε από την ψηφιοποίηση αυτή. Ευχαριστώ. Duda, και Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, η χώρα σας είναι από τους ηγέτες της ψηφιακές εξελίξεις. Έχω κάποιες ερωτήσεις επ' αυτού. Πώς θα συνεργαστείτε με τους συναδέλφους σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονιζόμενοι για να άρετε τους, τους φραγμούς, για να πετύχετε τους στόχους. Τι κριτήρια θα χρησιμοποιήσετε για να αξιολογήσετε ποια δράση θα πρέπει να δρομολογηθεί. Θα δεσμευτείτε να χρησιμοποιείτε περισσότερο τις αξιολογήσεις συνεπιών για να αποτιμήσετε τα μέτρα εκείνα που πιθανόν θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και να βασίζετε επ' αυτού τις προτάσεις σας. Και τέλος, εάν μπορούσατε να επιλέξετε ένα μέτρο και μόνο που θεωρείτε ότι θα παράγει τη μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη για την ενιαία ψηφιακή αγορά, ποιο θα ήταν αυτό. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ευχαριστώ για την ερώτηση ή τις ερωτήσεις μάλλον. Όπως γνωρίζουμε, πολλές ομάδες προβληματισμού πριν από 5-10 χρόνια ε, πρότειναν να οργανωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσκη διαφόρων συστάδων ομαδοποίησεων θεμάτων. Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο πρόεδρος, ο επόμενος, αποφάσισε να διοργανώσει τη δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει τέτοιων συστάδων και οι αντιπρόεδροι θα κινούνται βάσει των οδηγιών του Προέδρου και θα συντονίζουν διάφορους τομείς πολιτικής. Περισσότερο συντονισμός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν κάτι που χρειαζόταν ήδη εδώ και κάποια χρόνια και χρειάζεται ακόμα περισσότερο τώρα κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών σεμιναρίων που είχαν διοργανωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποιοι γενικοί διευθυντές που συμμετείχαν είπαν «Κοιτάξτε, ήδη δουλεύει το πράγμα, εδώ είμαστε, καθόμαστε και συζητάμε τα ίδια ζητήματα. Προστασία των δεδομένων, εμπιστοσύνη. ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών κλπ. κλπ. Δεν συνέβαινε όμως τόσο συχνά. Διάφοροι ειδικοί από διάφορες γενικές διευθύνσεις να κάθονται μαζί να συζητάνε τα ίδια θέματα. Αξιολόγηση συνέπειων. Ναι, αυτή είναι η βάση. όλες οι προτάσεις που ετοιμάζαμε ε, συνεπάγονται και την προετοιμασία αξιολογής συνεπειών. Ζητώ συγγνώμη γιατί έληξε ο χρόνος στη διάθεσή μου. Και το θέμα των δεξιοτήτων. Οι ψηφιακές δεξιότητες των παιδιών μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Κυρία Σοραντσόβα από την Άλντε της Επιτροπής ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ Προέδρε, αγαπητέ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Όπως βλέπετε υπάρχει μεγάλη υποστήριξη σε αυτό που είπατε. Πράγματι δέχονται τη γη της Εστονία ε, στις ε, δημόσιες και τις εμπορικές ε, ψηφιακές υπηρεσίες και τις ψηφιακές υπηρεσίες. Θέλουμε όμως να έχουμε, δεν έχουμε μια αγορά σε αυτό το βαθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κατακαιρματισμένη σε 28 εθνικές αγορές και υπάρχει προστατευτισμό σε κάθε χώρα. Είπατε επίση ότι η Εστονία δεν είναι τέλεια και δεν μπορεί να διδάξει τους άλλους. Από τη δική σας όμως εθνική εμπειρία και τη συνεργασία σας με άλλα ποια εθνικά μέτρα θεωρείτε ότι είναι επιτυχή και πώς μπορείτε αυτά να τα φέρετε στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην αγορά της Ένωσης, είσαστε υπέρ συντονισμού εθνικών προσπαθειών ή θέλετε πιο εναρμονισμένα συστήματα που θα, είναι, θα καλύπτουν όλη την Ευρώπη. Απάντηση, ευχαριστώ. Όπως τα περιγράψατε έχουν τα πράγματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε 28 ε, διαφορετικές νομοθεσίες για τα ψηφιακά θέματα. 28 έξοχες νομοθεσίες αλλά διαφορετικές για την ηλεκτρονική τεχνολογία που καλύπτουν τα ψηφιακά θέματα. Και αυτές οι έξοχες νομοθεσίες δημιουργούν φραγμούς μεταξύ των κρατών μελών. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια πραγματική ενιαία ψηφιακή αγορά δεν θέλω να αναφερθώ εκτενώς στα παραδείγματα της Εστονίας. Σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούμε να βρούμε πολύ καλά παραδείγματα που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν παράδειγμα για άλλους. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ήταν, όχι, μάλλον είναι επιτυχής στην Δανία και τώρα γνωρίζω ότι αποτελεί επιτυχία και στην Ισπανία και στην Ιταλία καθώς και στην Φιλανδία. Τώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποστηρίξουμε τη διάδοση των βελτίστων πρακτικών και να βρούμε καλές ηλεκτρονικές λύσεις που αφορούν το διαδίκτυο. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζονται κοινέ προδιαγραφές για ηλεκτρονική τιμολόγηση. Έχει δρομολογηθεί η θέσπιση κανόνων, κοινών κανόνων και ελπίζουμε ότι τελικά θα χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική τιμολόγηση σε όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Κυρία Βερζιά από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για την ΚΟΕ. ευχαριστώ. Είναι σαφή η θητεία σας το να μεταμορφωθεί η Ευρώπη σε παγκόσμιο ηγέτη στις τηλεπικοινίε και τον ψηφιακό κόσμο, ώστε να επιτρέψουμε την βελτιστοποίηση τη χρήση του. Θέλετε να προωθήσετε τη χρήση του ψηφιακού και σε σχέση με την οικονομία, μόλι το ακούσαμε. Εμείς στην ΚΟΕ δεν πιστεύουμε στις αρετές τη αγορά για τη ρύθμιση των προβλημάτων. Ξέρουμε ότι έχει πλέον κτήματα ο ψηφιακό κόσμο, όχι όμω χωρί κινδύνου, ιδιαίτερα για την ασφάλεια των πολιτών όπω και των επιχειρήσεων εξάλλου, η προστασία τη θετική ζωή και των δεδομένων. Εμεί λοιπόν στη ΛΥΜΠΕ, μετά από τι εμπειρίε που είχαμε τι ΗΠΑ, ε, θα θέλαμε να αντιδράσουμε. Και ο κίνδυνο συμπεριλαμβανομένων και των επιθέσεων προέρχεται από τι ε, χώρε επίση. Πέρα από αυτές τις γενικότητες που μας αναφέρατε, ποια συγκεκριμένα μέτρα μας προτείνετε, πέραν δηλαδή από την εφαρμογή του πακέτου για την προστασία των δεδομένων, ποιες προτάσεις ε, για την αναθεώρηση του Safe Harbor, για τις τηλεπικοινωνίες και για τις συμφωνίες με τρίτες χώρες και ιδιαίτερα με τις πολιτείες, μας προτείνεται. Thank you. Ευχαριστώ. Καταρχάς για την ενιαία αγορά. Ξέρετε ότι εμείς δεν πιστεύουμε στις αγορές. Ως φιλελεύθερος εγώ πιστεύω στις αγορές. Αλλά δεν νομίζω ότι η αγορά από μόνη της μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Η αγορά λοιπόν μπορεί ας πούμε να προστατεύσει το πιο ασθενές τμήμα της ε, κοινωνίας. Αντί για το κοινοβούλιο. Όχι, εμείς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πιστεύω και ως φιλελεύθερος στα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει να προστατεύουμε την ειδική ζωή των πολιτών και είναι υποχρεωτική η προστασία των δεδομένων όταν μιλάμε για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Καταρχάς λοιπόν θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το πακέτο προστασίας δεδομένων στο εσωτερικό της Ένωσης, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τον Γενάρη, ο πρόεδρος τον είπα, ο Μπαράκ Ομπάμα, έκανε μια θαυμάσια ομιλία είπε ότι όλα τα δεδομένα άσχετα με το αν είναι αμερικανικά αυτά τα δεδομένα Αμερικανών ή άλλων θα πρέπει να προστατεύονται επίσης όρις. Ήταν λοιπόν μια πολύ ισχυρή πολιτική δήλωση αυτή. Αναμένουμε λοιπόν κάτι αντίστοιχο για να μέναμε κατά αντίστοιχο τα τελευταία δέκα χρόνια. Αλλά αυτή η δήλωση τα 10 τελευταία χρόνια δεν προήλθε από τις πολιτείες. Τώρα αντίθετα βλέπουμε να υπάρχει μια, έτσι, μια πολιτική βούληση και θα δούμε κατά πόσο οι Αμερικανοί πραγματικά μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα λόγια και να τα κάνουν πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, πρέπει να σας πενθυμίσω το θέμα του χρόνου, διότι θα αργήσουμε. Η Τζούλια Ρέντα από την Επιτροπή Ίνκο. Μπροστά αριστερά. Κύριε Επίτροπε, υποψήφιε Επίτροπε, εδώ είμαι. Ο κόσμος ζητάει περισσότερη συμμετοχή στα θέματα που αφορούν το ίντερνετ. Αυτό το είδαμε, ας πούμε, στις διεθνείς διαδηλώσεις κατά του ΆΚΤΑ, που οδήγησαν στην ήττα του εδώ στο Κοινοβούλιο και από τον πολύ μεγάλο αριθμό απαντήσεων στις διαβουλεύσεις για τα πνευματικά δικαιώματα που οργάνωσε η Κομισιόν. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και ερωτήσεις που με ρώτησαν εμένα οι χρήστες του Ιντερνετ για να σας μεταφέρω και δυστυχώς δεν έχω χρόνο να τα θέσω όλα άμεσα. Σας ρωτάω αντίθετα ένα απλό ερώτημα. Είστε διατεθειμένος να εισέλθετε σε διάλογο με την ε, κοινότητα του ίντερνετ να υπάρχει δηλαδή μια επίσημη online ακρόαση όπου ο κόσμος θα μπορούσε να θέσει ερωτήματα. Θέλετε και μπορείτε να κάνετε αυτό το τολμηρό βήμα πριν αναλάβετε τη, τα καθήκοντά σας. Ε, δέχεστε κάτι τέτοιο ναι ή όχι. Ευχαριστώ για το ερώτημα. Το συζητήσαμε νωρίτερα. Η απάντηση είναι ναι. Δέχομαι, δέχομαι. Και είμαι έτοιμος να συμμετάσχω σε ακροάσεις online με συζητήσεις με τους πολίτες μας. Αναφερθήκατε στην άκτα. Εγώ ίδιος προσωπικά υποστήριξα την άκτα γιατί από ό,τι κατάλαβα εγώ η βασική του άκτα ήταν καλή. Δηλαδή το να θεσπίσουμε κοινέ προδιαγραφές σχετικά με την προστασία των πραγματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και στις τρεις χώρες. Όμως η διαδικασία ήταν πραγματικά απέσια. Δεν ήταν καθόλου περιληπτική και γι' αυτό ακριβώς το λόγο τα αποτελέσματα ήταν αυτά που ήταν. Οπότε θα πρέπει να μάθουμε ακριβώς από την υπόθεση της άκτα. Θα πρέπει να δράσουμε με ένα πιο περιληπτικό τρόπο Ευχαριστώ. Diane James. Diane James από το EFTD, πάντοτε στην ΕΜΚΟ. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. My apologies. Ζητώ συγγνώμη, λέει Μιλίτα. Να ξαναρχίσουμε το ρολόι σας, παρακαλώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Δηλώσατε ότι η ανάπτυξη τη ψυχική οικονομία έχει τεράστια σημασία. Όμω ο μεγαλύτερο κίνδυνο είναι αυτός που εμφανίστηκε Μάρτι φέτος που συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του Ετού. ήταν η άρνηση υπαρχή υπηρεσία μετά από, ιδιαίτερα από την κρίση στην Ουκρανία σε πάρα πολλέ περιοχές. Μπορείτε να μας δώσετε κάποιε διαβεβαιώσει σε σχέση με το ποιε προτεραιότητες θα δώσετε ακριβώς αυτό το τομέα, ποιες, ποιους πόρους θα αφιερώσετε εκεί και ποιο θα είναι το επίπεδο αυτού του θέματος στην ημερήσια διάταξή σας νωρίς στη θητεία σας. Μπορείτε να μας δώσετε λεπτομέρειες. Ναι, από ό,τι κατάλαβα, μιλάμε για την προστασία των καταναλωτών. Κατά την άποψή μου, μεταξύ όλων αυτών των ψηφιακών λύσεων. Η ενιαία ψηφιακή αγορά θα πρέπει να παραμείνει στο πλευρό των καταναλωτών. Εάν οι καταναλωτές δεν, δεν προστατεύονται συγγνώμη, σωστά, εάν οι πολίτες μας, οι καταναλωτές δεν έχουν εμπιστοσύνη σε αυτές τις καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, δεν θα τις χρησιμοποιήσουν ποτέ προφανώς. Οπότε, όπως είπα στην αρχική μου ομιλία, οι πολίτες, ο κόσμος, νομίζω αποτελούν το σημείο κίνηση σε όλες τις διαδικασίες. Και η εμπιστοσύνη αποτελεί τη βάση για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες. Οπότε τώρα έχουμε πολλές καλές πρωτοβουλίες που είμαι βέβαιος ότι θα βοηθήσουν να οικοδομηθεί αυτή η εμπιστοσύνη όπως το πακέτο για την προστασία δεδομένων, η ενιαία αγορά ψηφιακή και πάλι η προστασία των καταναλωτών βρίσκεται σε πολύ ψηλό επίπεδο χάρη σε αυτό το πακέτο. Μετά, κοινό ευρωπαϊκό νόμο για την προστασία των καταναλωτών. Και πάλι αυτό θα αποτελεί μια εναλλακτική, αλλά σε τελική ανάλυση θα βοηθήσει τους πελάτες και βεβαίω τι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσει. Οπότε οι καταναλωτέ θα πρέπει να αποτελούσουν πραγματικά το επίκεντρο όλων αυτών των διαδικασιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Τονζίνσκη από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγορά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Υποψήφια Επίτροπε η ψηφιακή αγορά, η ενιαία ψηφιακή αγορά έχει σαν στόχο να διευρύνει και να διευκολύνει τι συναλλαγέ μεταξύ των διαφόρων χωρών τη Ένωση. Το καταλάβαμε καλά, γνωρίζουμε και πόσο σημαντικό είναι αυτό. Φιλοδοξία είναι να δημιουργηθούν ευκαιρίε για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, διευκολύνοντα την πρόσβασή του σε εθνικέ αγορέ σε διακοινωτικό επίπεδο. Παρομοίω, ε, θα ε, ευνοηθεί η παραγωγή, οι αγορέ, ο εφοδιασμό και άλλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων προ χώρε όπου έχουν χαμηλότερο κόστο παραγωγή ακόμα και εντό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Κυρίως προς χώρες της Ανατολής όπου το κόστος το εργατικό είναι πολύ πιο χαμηλό. Δεν φοβόσαστε λοιπόν ότι βγάζοντας τελευταίους φραγμούς που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της ψηφιακής ενίας αγοράς ότι το δραματικό φαινόμενο της μεταγκατάστασης που έχει βλάψει πολύ το γαλλικό λαό μήπως εντατικοποιηθεί περαιτέρω. Thank you. Σας ευχαριστώ. Βέβαια, η ψηφιακή ενιαία αγορά θα στηρίξει κυρίως τις μικρές και μεσαίου μεγέθους εταιρείες. Η ενιαία ψηφιακή αγορά θα διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γνωρίζουμε το, για τον νομοθεσία την κοινή την ευρωπαϊκή για τις πωλήσει που θα βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις να πολλούν στο διαδίκτυο ή να πολλούν σε άλλες χώρες. Οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να αντιμετωπίζουν 28 διαφορετικές ε, νομοθεσίες. Για μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις όμως είναι αδύνατο. Δεν μπορούν να γνωρίζουν τις λεπτομέρειες των εθνικών νομοθεσιών. Όπως είπα και στην αρχή, αυτός ο κατακαιρματισμός θα σταματήσει την ανάπτυξη της επιχείρησής τους. Η ενιαία ψηφιακή αγορά θα δημιουργήσει συνθήκες για την ανάπτυξη όλων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ανεξάρτητα από το που βρίσκονται στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι η αυτή ψηφιακή αγορά θα οδηγήσει σε μεταγκατάσταση προς τις ανατολικές χώρες της Ευρώπης. Όπως είπα και προηγουμένως, η δημιουργικότητα, οι τέχνες, η γνώση που συμπεριλαμβάνεται στα προϊόντα, το ποσοστό όλων αυτών των στοιχείων στα προϊόντα αυξάνεται με ταχύ ρυθμό. Η γνώση, οι τέχνες. Δεν νομίζω ότι θα μετεγκατασταθούν μαζί με την ψηφιακή αγορά προς την Ανατολική Ευρώπη. Αυτός ήταν ο πρώτος γύρος των ερωτήσεων των πολιτικών ομάδων. Θα είμαι πιο αυστηρή όσον αφορά το χρονόμετρο και θα σας διακόπτω, λέει ο Πρόεδρος. Αν, ακόμα και αν κάνετε 5 δευτερόλεπτα παραπάνω και τον Επίτροπο όταν ξεπεράσει το χρόνο του κατά 10 δευτερόλεπτα. Thun und Holstein του ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρωθυπουργέ, λέει Μιλήτρια. Κάνουμε λόγο για τον κατακαιρματισμό της αγοράς. 28 ξεχωριστά κομμάτια σε αυτή την αγορά. Αυτό που είναι σημαντικό είναι οι συναλλαγές στο διαδίκτυο ηλεκτρονικά. Έχουμε 28 διαφορετικά συστήματα και τις ταχυδρομικές υπηρεσίες σε αυτές τις χώρες που τροχοπεδούν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ερώτησή μου, θα καταφέρετε να εμπλακείτε για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Τι στοχεύετε να πράξετε ώστε να υπάρξει μία ενιαία αταχυδρομική αγορά ώστε να μπορεί να αγοράζει κανείς και να πωλεί μέσω του διαδικτύου. Η κυρία Κρότς είπε ότι μέχρι το 2016 δεν θα έχουμε τις επιπτώσεις της, ε, των τελών περιαγωγής. Τι θα γίνει σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών, θα δώσετε μάχη πέρα αυτών. Ο κύριος Σφάμπ ανέφερε κάτι που θέλω να το τονίσω κι εγώ. Θέλουμε μια ενιαία εσωτερική αγορά ένα ενιαίο πλαίσιο και όχι 28 διαφορετικά καθεστώτα. Πώς θα πείσετε τους συναδέλφους σας στο Συμβούλιο για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Thank God. Yeah. Ναι. I'm going to make it work, Yeah, question. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Συμφωνώ μαζί σας. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες καμιά φορά εμποδίζουν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Αν πρέπει να πληρώσει κανείς πέντε φορές παραπάνω για τέλη αποστολής, δεν θα τα παραδώσει αυτά τα αγαθά σε άλλη χώρα, διότι σκοτώνει την επιχείρησή σου και δημιουργεί προβλήματα και για τους πελάτες. Αν έχουμε τη βάση στο Λονδίνο, η παράδοση στη Γλασκόβη είναι πολύ φθηνότερη από τις Βρυξέλλες. Μικρή, μικρότερη απόσταση Λονδίνο-Βρυξέλλες βέβαια. Υπάρχουν σύνορα που χωρίζουν και διαιρούν, μας διαιρούν. Όπως γνωρίζουμε όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση χωρίς σύνορα. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Η οδηγία για τις καθολικές υπηρεσίες. Πρέπει να δούμε ακριβώς τι θα καλύπτει το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας. Πρέπει να θέσουμε κανόνες. Πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι ισότιμα βάσει των κανόνων. Να μην πληρώνει ο κόσμος περισσότερα μόνο και μόνο γιατί υπάρχουν σύνορα. Αναλαμβάνω τη δέσμευση να βρω καλές λύσεις για τους πελάτες και είμαι σίγουρος ότι θα λυθούν και τα προβλήματα των ταχυδρομικών ε, υπηρεσιών. Εβελίν Γκέπχαρτ, σοσιαλιστές. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε... Σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, εσείς είπατε ότι μια ολιστική συνολική προσέγγιση θέλετε να έχετε και θα συνεργαστείτε στενά με τους άλλους επιτρόπους μεταξύ άλλων και με την κυρία Γιούροβα, τον κύριο Έτιγκερ. Πώς θα το κάνετε αυτό τελείως συγκεκριμένα και χειροπιαστά. Αναφέρατε και τους γενικούς διευθυντές, αλλά εμένα θα με ενδιέφερε πώς μεταξύ των επιτρόπων μπορεί να διασφαλιστεί και να διαμορφωθεί μια τέτοια συνεργασία. Είπατε ότι τους πολίτες, τους καταναλωτές θα τους θέσετε στο προσκήνιο, στην πρώτη γραμμή. Το χαιρετίζω αυτό, αλλά πώς θα το κάνετε, με ποιον τρόπο θα επιτευχθεί αυτό. Εκτός τούτων είπατε επιπλέον ότι θέλετε να μεριμνήσετε όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι πολίτες στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε αυτές τις δυνατότητες και είναι πολύ σωστό αυτό <clears throat> και για τους καταναλωτές και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδιαίτερη σπουδαιότητα για αυτές. Με ποιο τρόπο θα το κάνετε αυτό. Πώς θα υποστηρίξετε τα κράτη-μέλη για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πώς θα συνεργαστούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αντιπρόεδροι κυρίως και ο πρόεδρος. Ήμουνα πρωθυπουργός τη Εστονίας τα τελευταία 9 χρόνια. Πάντα είχαμε κυβερνήσει συνασπισμού στη χώρα. Και προϋποθέσεις για το συνασπισμό είναι η συνένεση αν ξεκινήσει κανείς με ψηφοφορίες, αμέσως πρέπει να βρει άλλους ε, εταίρους για, την, για το συνασπισμό. Έχω γεράσει πια για να αλλάξω συμπεριφορά. Θα συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ρόλος των αντιπροέδρων είναι να κατευθύνουν και να συντονίζουν. ρόλος των επιτρόπων είναι κάπως διαφορετικός. Να οργανώνουν και να διαχειρίζονται. Ο ρόλος του αντιπροέδρου είναι πιο οριζόντιος. Ο ρόλος του επιτρόπου είναι πιο κάθετος. Συμπληρωματική είναι αυτή η ρόλη. Και θα ήθελα να πω ότι και οι δύο ρόλοι χρειάζονται. Ευχαριστώ. Τίμωθη Κέρκχοπ e ε, για το ECR από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Υποψήφια επίτροπε, η ερώτησή μου αφορά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για το δικαίωμα να λησμονείται κάτι. Πώς θα διαμορφώνεται η πολιτική στην Ευρώπη, κυρίως όσον αφορά την καταπολέμηση του εγκλήματος και των επιχειρήσεων και όσον αφού τη διαγραφή, την παραγραφή και πώς όλα αυτά ταιριάζουν με την ελευθερία της έκφρασης και διάφορα δικαιώματα ιδιωτική ζωή, ζωής και η παραγραφή των αδικημάτων, η δικαίωμα όλων ή αποτελεί ε, μία εξαίρεση για τους λίγους. Thank you very much for this question. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Από ό,τι καταλαβαίνω, οι πολιτικοί δεν χρειάζεται να θεωρούν ότι θα λησμονηθούν τα λόγια τους. Όταν μιλάμε για το δικαίωμα να λησμονηθεί κανείς, να παραγραφεί κάτι, δεν μιλάμε για πολιτικούς. Θα τους θυμόμαστε και αυτό είναι καλό για τη δημοκρατία. Τι είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεν είπε ότι όλοι έχουν το δικαίωμα αυτό της παραγραφής ή της διαγραφής. Αλλά ήδη πριν από 10 και περισσότερα χρόνια στην νομοθεσία μας αναφερόταν ότι η προστασία των δεδομένων είναι κάτι που χρειάζεται για συγκεκριμένη προσωπική χρήση και για ορισμένο χρονικό διάστημα. Και μετά από αυτό δεν επιτρέπεται να διατηρούνται ακόμα αυτά τα στοιχεία. Πρέπει να διαγράφονται. Νομίζω ότι το δικαίωμα αυτό της διαγραφής πρέπει να παραμένει ως εξαίρεση. Το πραγματικό θέμα είναι πώς να βρεθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ της ελευθερίας της έκφρασης και της προστασίας της ιδιωτικής ζωής όλων. Αυτό θα εξετάζεται κατά περίπτωση και δεν είναι κανόνας που αφορά τους πολιτικούς της ΑΛΤΕ από την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Αν έχετε την καλοσύνη γυρίστε εδώ πίσω σας. Θέλουμε όλη την ψηφιακή ανάπτυξη, το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να δώσει πολλά και καινούργια ενδιαφέροντα πράγματα στους καταναλωτές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε δημιουργικό επίπεδο. Αυτό το ηλεκτρονικό, το ψηφιακό εμπόριο που θα αναπτυχθεί συνεπάγεται και νέες εμπορικές πρακτικές που είναι επικρίσιμες και καμιά φορά αθέμητες, όπως οι κρυφές διαφημίσεις ε, ή ε, ψευδείς διαφημίσεις ή συγκρίσεις διαφόρων προϊόντων, καταχρηστική χρήση προσωπικών δεδομένων. Λοιπόν, στην Ένωση υπάρχει μια οδηγία που είναι κατά το θέμι των αθέμητων πρακτικών, που είναι βασικό εργαλείο για να προστατευτεί ο καταναλωτής. Αρκεί την ψηφιακή εποχή αυτό χρειάζεται κάποιο άλλο εργαλείο νομοθετικό για να ενισχυθεί κατά πολέμηση των νέων πρακτικών. Και αν υπάρχει κάτι τέτοιο, ποια πρακτική, πώς θα βελτιώσετε τα πράγματα με συγκεκριμένο όμως τρόπο. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Φτάνει. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει. Οπότε εμεί θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να προστατεύσουμε τους πολίτες μας, για να προστατεύσουμε τους πελάτες μας. Ηλεκτρονικό εμπόριο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν είναι κάτι το φανταχτερό και εφημερό. Θα παραμείνει για πολύ καιρό μαζί μας. Τώρα το ηλεκτρονικό εμπόριο αντιπροσωπεύει το 5% του λιανικού. Όμως είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα αυξηθεί το μερίδιο του ηλεκτρονικού εμπορίου ταχύτατα και εμείς θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις και τους πελάτες περιβάλλον για το ηλεκτρονικό εμπόριο. αυτή η δυναμική τιμολόγηση, dynamic pricing, είναι κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό. Αν θα πρέπει να πληρώσετε ψηλότερε τιμέ επειδή έχετε επιθέσει ε, στην ηλεκτρονική σα διεύθυνση, αυτό είναι καθόλου ευχάριστο. Βεβαίω, αν υπάρξουν προτάσεις, αν ας πούμε προτείνουν προτείνουν έτσι προϊόντα όπως μουσική που θα σας αρέσει ταυτόχρονα ας πούμε με την κυβερνοεπίθεση εντάξει ίσως να το δεχόμασταν αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν με νοιάζουν τα θέματα τα ιδιωτικότητα από τη στιγμή που δεν πληρώνω. Όμω αυτό έχει και ένα τίμημα. Και ε, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και εμάς στο Κοινοβούλιο, αλλά και, και εμάς στην Επιτροπή, αλλά και στο Κοινοβούλιο. Κονέλη Άντς για την ΓΚΟΕ. Εδώ αριστερά σας. Θα ήθελα να σας διατυπώσω μια ερώτηση όπως την έθεσα ήδη στο παρελθόν προς τον κύριο Έτιγκερ που δεν την ε, απάντησε. Πρόκειται για την ε, ε, πληροφορική και την ασφάλεια της πληροφορικής και της ηλεκτρονικής βιομηχανίας. Δουλειά σας είναι να επικαιροποιηθεί και να εξυγχρονιστεί αυτός ο τομέας, είναι σαφές και για τις ε, μαζικές ε, κατασκοπίες, τη μαζική κατασκοπία βάρος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποβληθεί μια ολόκληρη σειρά προτάσεων και έχουν ζητηθεί να υλοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα απάντηση από αυτού από εσά. Πρώτη ερώτηση. Θα υποβάλλετε προτάσεις εσείς ο ίδιος ώστε πόρτες και παράθυρα να κλείσουν ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται με ασφάλεια περισσότερο λογισμικό. Δεύτερον, θα προωθήσετε με σθένος την ηλεκτρονική βιομηχανία συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών εγκεφάλων, υπολογιστών και της κρυπτογράφησης ε, θα προωθήσετε το τομέα αυτό της IT, της ηλεκτρονικής τεχνολογίας πληροφοριών και πώς θα το κάνετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο τζίρο πλασιάζεται κάθε δύο χρόνια. Κωδικοποίηση. Η κωδικοποίηση, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. κωδικοποίηση. Στην Ένωση προωθούμε το ανοιχτό λογισμικό. Οπότε δεν χρειάζεται να αρχίσουμε από το μηδέν. Ξέρω από την θητεία μου ως πρωθυπουργός στη χώρα μου βέβαια που γνωρίζω πολύ καλά είχαμε την πρακτική ως εξής. Εάν αυτό το λογισμικό στη χώρα μας που δημιουργήθηκε στη χώρα μας δέχεται κοντήλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε αυτό το λογισμικό θα πρέπει να είναι ανοιχτό και για άλλους χρήστες. Αν εμείς θέλουμε να έχουμε λύσει στα μέτρα μας, τότε νομίζω ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Οπότε η Ένωση, η Κομισιόν από την άποψη αυτή νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουν ακριβώς την χρήση του ανοιχτού λογισμικού και ήδη το πράττουν. Βεβαίως εγώ σχεδιάζω βεβαίως και προτίθεμαι να υποστηρίξω κάθε εξέλιξη σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Περάσαμε το 1 τέταρτο της διαδρομής. Τζούλια Ρέντα από τους Πράσινους ξανά. Yes, me again. Um, εγώ και πάλι, ναι. Με χαρά άκουσα στην αρχική σας δήλωση ότι θέλετε να περιλάβετε την ουδετερότητα στον νόμο, στην νομοθεσία. Το θέμα όμως πώς προσδιορίζετε την κυβερνητική, την ψηφιακή ουδετερότητα. Είχαμε τον πακέτο στο Κοινοβούλιο που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα και πρότεινε κάποιες λύσεις, κάποιες ε, προτάσεις. Συμφωνείτε με τον ορισμό του Κοινοβουλίου όσον αφορά την ε, ουδετερότητα. Προτίθεστε να την αθετήσετε. Και βεβαίως αυτό το θέμα της ουδετερότητας σχετίζεται άμεσα με άλλα ζητήματα όπως η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλα. Τι γίνεται λοιπόν με την ουδετερότητα όσον αφορά την αναθεώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων, προστασία των δεδομένων κλπ. Είστε διατεθειμένος να διασφαλίσετε την συνάφεια της υπάρχουσας νομοθεσίας με την αρχή της ουδετερότητας της ψηφιακής. Uh, net neutrality is a really important Ευχαριστώ. Ναι, το θέμα αυτής της είναι σημαντικό και νομίζω ότι όλοι οι ευρωβουλευτές μπορούν να είναι υπερήφανοι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αρχή της Ιντερνετικής ιδιωτερότητας ρυθμίζεται σε επίπεδο νομοθεσίας. Μιλάω για το πακέτο ενιαίας αγοράς των τηλεπικοινωνιών. όλη η ανταλλαγή δεδομένων στο ίντερνετ θα πρέπει να είναι αντικείμενο ίσης μεταχείρισης. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να κάνει καταχρήσεις, ιδιαίτερα της δεσπόζουσας θέσης, του στην αγορά ή της θέσης του ως φύλακα. Όπως ξέρουμε, σε κάποιες μηχανές αναζήτησης δεν μπορούμε να, να συστήσουμε να μιλήσουμε για ουδετερότητα ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες. Πολύ συχνά είναι απολύτως αδύνατον να βρει κανείς προβολή και να εμφανίζεται σε αυτές τις μηχανές αναζήτησης. Οπότε, αν δεν μπορείτε να έχετε έτσι προβολή στις μηχανές ε, αναζήτησης, δεν μπορείτε και να πουλήσετε τα προϊόντα σας. Οπότε δεν έχει νόημα και να παράγεις κάτι. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν η Ιντερνετική αποτελεί μια βασική αρχή, μια σημαντική αρχή για τους πολίτες μας αλλά και για τις επιχειρήσεις μας. Τώρα για την ταχύτητα. Η υψηλότερη τιμή για υψηλότερες ταχύτητες είναι κάτι αποδεκτό. Όχι όμως εις βάρος των υπολείπων. Όχι εις βάρος αυτών των οποίων η ταχύτητα ήδη είναι χαμηλή. Αποκλείεται αυτό. Ευχαριστώ from the EFDD Diane James από το FTD και πάλι. Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονική πρόσβαση. Υποψήφια επίτροπε σε όλου του τομεί αποτελούν ενδεχομένω του τομεί με τη μεγαλύτερη αύξηση και ανάπτυξη ε, στι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε. Και το είχαμε συζητήσει και για το λιανικό εδώ στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, η πρόσβαση σε ίντερνετ υψηλή ταχύτητα είναι κάτι το άνισο και αυτό ενδεχομένως δημιουργεί προβλήματα. Δημιουργεί προβλήματα όσον αφορά τις προσφορέ, την αντιμετώπιση των μονοπωλίων, αφορά όσον αφορά τα συμφέροντα κρατικών τηλεπικοινωνικών οργανισμών στην Ένωση. Μπορείτε να μα δώσετε κάποια έτσι ιδέα για το πώς θα αντιμετωπίσετε τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ αυτών που βρίσκονται σε αυτού του τομεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δική σα θέση Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω αναφερθήκατε και στην ηλεκτρονική υγεία παλαιότερα. Όταν μιλάμε για τα θέματα ταχύτητα στο ίντερνετ, θα πρέπει να υπάρχει επίσης και το περιθώριο εξαιρέσεων και η υγεία, το μέσο υγείας είναι μία από αυτές τις πιθανές εξαιρέσεις. Εάν το ερώτημα είναι σχετικό με τις ανθρώπινες ζωές, αν περί αυτού δηλαδή έχουμε να κάνουμε, τότε αυτές οι πληροφορίες, οι πληροφορίες που αφορούν την ηλεκτρονική υγεία, προσωπικά δεδομένα υγείας κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα όταν αυτά τα δεδομένα κινούνται στο ίντερνετ. Έχουμε πάρα πολλά συστήματα ηλεκτρονικά υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερθήκατε προηγουμένως στα συμφέροντα στις, ε, στους, στους οργανισμούς τηλεπικοινωνιών. Να σας μιλήσω για τα συμφέροντα που αφορούν τα νοσοκομεία. Εμείς εδώ στην στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είμαστε πολύ περήφανοι για την ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών. Όμως πόσο σοβαρά μπορούμε να μιλήσουμε για την ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών όταν σε κάποιες χώρες οι ασθενείς δεν έχουν καν δικαίωμα να λάβουν αντίγραφο του προσωπικού ιατρικού φακέλου. Πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία για να ε, ρωτήσουν, πούμε να ζητήσουν την άποψη κι άλλου γιατρού τη δεύτερη γνώμη που λέμε. Οπότε βεβαίως υπάρχουν αυτά τα συμφέροντα και εγώ δεν θέλω μόνο να ασχοληθώ με ένα τομέα, τομέα μόνο των τηλεπικοινωνιών γιατί τα συμφέροντα υπάρχουν παντού σε όλους τους τομείς. Ευχαριστώ. Πελέμψικη από τη Λίμπε, Έχει μέσα το γεγραμμένων. γραμμένον. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίτροπε. Πρώτον, η εξέλιξη και ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούσαμε πολλές τοποθετήσεις. Ένας πραγματικός ε, ρόλος κλειδιού θα μπορούσε να είναι η φορολογική ελάφρυνση και διευκόλυνση, τουλάχιστον όσο αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ερώτηση, πώς μπορείτε εσείς ε, να χρησιμοποιήσετε και να δημιουργήσετε αυτό το μέσο, ώστε να υπάρξει επαναστατική δράση και εφαρμογή μέσω αυτού του μέσου στην ψηφιακή αγορά και σε σχέση με τις παράνομες επιθέσεις στα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εις βάρος των πολιτών. Ερώτηση. Πώς βλέπετε την αντίδραση με βάση τη σκέψη σας όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν επανειλημμένα τέτοιες παράνομες επεμβάσεις καταχρηστικά εις βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Uh, Ψηφιακή ενιαία αγορά και οι φορολογικές απαλλαγές για ψηφιακά προϊόντα. Με τα λύπη μου λέγω ότι δεν υποστηρίζω τις μειώσεις φόρων και τις φοροαπαλλαγές Δεν είναι πολύ δύσκολο θέμα. Θα λάβουμε τις αποφάσεις στο σώμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει συνενέσεως. Είμαι έτοιμος για συνένεση. Κατάγομαι από μια χώρα όπου δεν είχαμε και δεν έχουμε τόσες πολλές μειώσεις φόρων και φοροαπαλλαγές και δεν υποστηρίζω τις φοροαπαλλαγές. Διότι το φορολογικό σύστημα, αν είναι διαφανές και απλό, κατανοεί όλα λαός πώς λειτουργεί και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν τους φόρους. Λένε είμαι ένας έντιμος φορολογούμενος, πληρώνω όλους μου τους φόρους, σύμφωνα με τον νόμο και δεν θα αναγνωρίζω γιατί η κυβέρνηση σπαταλάει τα χρήματά μου. Έτσι λειτουργεί. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους μηχανισμούς εποπτείας και να αναπτύξουμε νέες λύσεις για την ηλεκτρονική τεχνολογία. να δημιουργήσουμε περιβάλλον φιλικό προς επιχειρήσεις, να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις. Μπορούμε να βρούμε άλλα μέσα για να αναπτύξουμε την ψηφιακή βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τρίτος γύρος. Αντώνιο Λόπες Ιστουρίθ. White για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Αγαπητέ υποψήφια Πρόεδρε, έχουμε μια πιο εδρωμένη εσωτερική αγορά στο ψηφιακό που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 100% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για 520 δις ευρώ. Παρ' όλα αυτά, η τωρινή κατάσταση στον ψηφιακό κόσμο, στην ψηφιακή αγορά, παρουσιάζει κατακαιρματισμό. Έχουμε 28 αγορές, δηλαδή εθνικέ. Προηγουμένω μιλούσατε για τον κύριο Κατάουνεν, Κατάινεν. Ε, και εγώ θεωρώ τον εαυτό μου φιλελεύθερο. Εμεί κομμάστε στο σωστό κόμμα, το ΕΛΚ. Εσεί ε, βρίσκεστε σε ένα κόμμα κάπω πιο σοσιαλιστικό. Καμιά φορά πιο σοσιαλιστικό από το πρώτο κόμμα. Σα αυτό λοιπόν φιλελεύθερος. Θα υποστηρίξετε την ιδιωτική πρωτοβουλία σε αυτό το τομέα σε αυτόν τον τομέα της νέας ε, ψηφιακής αγοράς και ως φιλελεύθερος τι μέτρα θα υιοθετήσετε για την άστον των φραγμών που αποτρέπουν αυτό το, την υλοποίηση αυτού, τη, του, αυτού του της ψηφιακής αγοράς. Ευχαριστώ. Thank uh, Ευχαριστώ. Φυσικά έχουμε προτεραιότητα για τις επεμβάσεις, διότι το δημόσιο χρήμα είναι περιορισμένο. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε παντού δημόσια κονδύλια. Όμως, αναφέρατε επίσης τον Γύρκη Κατάινεν. Από κοινού πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε 300 δισεκατομμύρια ευρώ για να υποστηριχθεί η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα και τα κατανοώ, είναι πολύ σημαντικό να επενδυθούν αυτά τα κονδύλια με ένα πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και όταν γνωρίζουμε, αν γνωρίζουμε ότι ο ψηφιακός τομέας, η ψηφιακή οικονομία με μεγαλύτερη ταχύτητα αναπτύσσεται από ό,τι άλλοι παραδοσιακοί τομεί, τότε το σωστό πράγμα να πράξουμε είναι να επενδύσουμε στα ψηφιακά. Αυτό που πρέπει να δούμε τώρα, πρέπει να βρούμε πρόσθετα κονδύλια για επενδύσεις αυτή τη στιγμή. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Διότι το MFF ήταν ένας συμβιβασμός. Ήταν ένας αρκετά καλός συμβιβασμός κιόλας. Όμως, από την άλλη πλευρά, πιστεύω ότι δεν ήταν καλό, δεν, η ντροπή ήταν που δεν μπορέσαμε να προστατέψουμε κονδύλια που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τα ευρυζωνικά δίκτυα στην διασύνδεση των ευρωπαϊκών κρατών μεταξύ τους, Connecting Europe Facility. Αρχικά είχαμε 9 δισεκατομμύρια. Όμως για το, τα ευρυζωνικά και τις ψηφιακές ε, δυνατότητες ε, λύσεων, όμως συναθρηστικά για όλα τα κράτη-μέλη. Όλοι οι πρώην συνάδελφοί μου τι έκαναν. Ήταν όλοι υπέρ του να συνδεθούν τα κράτη μεταξύ τους, υπέρ του Connecting Europe. Όταν ξεκινήσαμε όμως να επιμερίζουμε τα κονδύλια αυτά, τα κεφάλαια αυτά, όλοι ήθελαν να πάρουν περισσότερα όσον αφορά τα εθνικά χαρτοφυλάκια, μεγαλύτερα και περισσότερα κονδύλια. Και τώρα πρέπει να δούμε και να διασφαλίσουμε άλλες πηγές, ώστε να υπάρξει πρόσθετη κεφαλαιοποίηση και διάθεση κονδυλίων για τη μόχλευση αυτών των επενδύσεων. Ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτή είναι μια ε, προοπτική. Αλλά Νομίζω τα κατάφεραμε σας στα πλαίσια του χρόνου. Για κονσάρι από τους Σοσιαδημοκράτες, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω φινλανδικά διότι κατανοούμε και οι δύο αμφότεροι την γλώσσα αυτή που ανήκει στην ίδια γλωσσική οικογένεια. Δεν απαντήσατε στην κυρία Γκέπαρντ. Πώς θα διασφαλίσετε ώστε οι περιοχές της υπαίθρου να έχουν ταχύτατη σύνδεση ψηφιακή. Οι ψηφιακές επενδύσεις στις υποδομές είναι το κλειδί εδώ νομίζω από πλευρά πλευράς σπουδαιότητας. Μέσα σε μια τέτοια δυνατότητα και προοπτική οι εταιρείε μπορούν να παράξουν και να είναι παραγωγικές. Συνήγαγα από τα όσα είπατε ότι είσαστε πρόθυμος τα 300 δισεκατομμύρια αυτά για το επενδυτικό πρόγραμμα του Juncker να λειτουργήσει και να συμπεριληφθεί και το ευρυζωνικό, τα ευρυζωνικά να συμπεριληφθούν και όλες οι άλλες επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την ψηφιακή επανάσταση στην Ευρώπη. Ένα άλλο πράγμα είναι το οποίο ελαφρά την καρδία αντιμετωπίζεται είναι τα θέματα τα φορολογικά. Όμως κύριε Άνσιπ, στο ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να εναρμονίσουμε τα πράγματα όσον αφορά τον ΦΠΑ και τα καθεστώτα ΦΠΑ. Διαφορετικά ποτέ δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τα πλαίσια και τα καθεστώτα ηλεκτρονικών ε, αγορών και συναλλαγών στο διαδίκτυο υπέρ των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Σα Σας äh, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πράγματι, κατανοώ τα φινλανδικά και μιλάω λίγα φινλανδικά, όχι όμως τόσο καλά και γι' αυτό θα μιλήσω αγγλικά. Και φυσικά είναι σωστό και πρέπει να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε μια ευκαιρία στο να δημιουργηθεί μια θετική πρόσβαση σε διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων και υπέρ εκείνων των πολιτών και για εκείνους τους πολίτες που ζουν στην Ήπεθρο και εκεί όπου οι δείκτες οι πληθυσμιακοί είναι χαμηλοί λόγω της αραιής κατοίκησης. Εκείνο το οποίο πρέπει να δούμε ότι το ε, πιο σημαντικό σε σχέση με το κόστος είναι η τελευταία σύνδεση και οι επενδύσεις που γίνονται από τις επιχειρήσεις γίνονται στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου ε, ο πληθυσμός είναι ε, υψηλής πυκνότητας. Εκεί υπάρχει υψηλό ποσοστό πληθυσμού στα αστικά κέντρα. Όπως όμως γνωρίζουμε η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα σήμερα, τουλάχιστον στην Ευρώπη για τους πολίτες της Ευρώπης και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να παράσχουμε ευκαιρίες ευκαιρίες για να χρησιμοποιείτε ε, το διαδίκτυο και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και από και για εκείνους που ζουν στην Ήπεθρο και στις ε, πιο απομακρυσμένες ε, περιοχές της Ήπεθρου. Το θέμα της φορολόγησης είναι πολύ ευρύτερο και είναι πολύ σημαντικότερο από ότι ε, είχα την ευκαιρία να απαντήσω στα 20 δευτερόλεπτα που είχα στη διάθεσή μου. Δεν είμαι όμως οπαδός του εναρμονισμού όσον αφορά τα ποσοστά ΦΠΑ στην Ευρώπη. Προτιμώ για παράδειγμα την εφαρμογή προτάσεων και προσεγγίσεων μιας ε, εταιρικής φορολόγησης ε, μέσα σε ένα παγιωμένο ή πιο ενιοποιημένο πλαίσιο που να μπορούν να υποφεληθούν οι εταιρείε και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ στα φινλανδικά. Ε, Κύριε Άνσιπ, έχω κάποια ανησυχία που αφορά την ψηφιοποίηση. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Η ψηφιοποίηση λοιπόν πράγματι εμπεριέχει πάρα πολλές δυνατότητες αλλά και απειλές όπως για την προστασία της ιδιωτικής ζωής όπως αναφέρατε. Ως γιατρός ε, γνωρίζω ότι αν θέλει να ανεβάσει κανείς το ιατρικό του ιστορικό στο διαδίκτυο δημιουργούνται προβλήματα. Θα μπορούσε όμως κανείς να αφεληθεί ε, να μπορούσα να χρησιμοποιήσω τα στοιχεία μου για την υγεία μου, για ηλεκτρονική υγεία, χρησιμοποιώντα τα έξυπνα τηλέφωνα κλπ. Το θέμα είναι τι θα κάνω με τα στοιχεία μου θα τα στείλω. Δεν είναι. Το διαδίκτυο βλέπετε πώ χρησιμοποιείται. Ε, και ιατρικά στοιχεία ίσω μπορεί να τριγυρνάνε στο διαδίκτυο. Πώ θα είναι ασφαλή αυτά, τι μέτρα μπορείτε να εφαρμόσετε ώστε να εμποδίσετε παράνομε δραστηριότητε κατά στοιχείων, ιατρικών στοιχείων που θα μπορούσαν παραδείγματο χάρη να, άμα γίνει κάποιο hacking, να μπορούν να διαδοθούν στο δημόσιο, στο κοινό, ανοιχτό κοινό, να αποκαλυφθούν ε, πληροφορίες ιδιωτικού χαρακτήρα. Thank Σας ευχαριστώ. Όπως είπα, σας ευχαριστώ. Όπως επανειλημμένα πολλές φορές ανέφερα σήμερα ήδη, η εμπιστοσύνη είναι βασικής αρχής ε, θέμα όταν κάνουμε λόγο για λύσεις στα ψηφιακά. Ιδιαίτερα όταν κάνουμε λόγο για τα θέματα υγείας, για την υγεία. Ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα. Ε, τότε λοιπόν πραγματικά η εμπιστοσύνη είναι υποχρεωτική, είναι επιτακτικού χαρακτήρα. Είναι επιταγή. Και γι' αυτό πρέπει να προστατέψουμε τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα με πολύ ασφαλή τρόπο, με τον πιο ασφαλή τρόπο. Η προστασία δεδομένων δεν είναι κάτι για ρυθμιστικές αρχές οι εταιρείε, οι επιχειρήσεις μας πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα της προστασίας δεδομένων. Επειδή ακριβώς υπάρχουν οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί προστασίας δεδομένων και ζητούν να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά προσέξτε, η προστασία δεδομένων είναι θέμα εμπιστοσύνης που θα βασίζεται σε θεμέλια εμπιστοσύνης. Είναι για τους ίδιους τους πολίτες μας ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Ένα κλίμα εμπιστοσύνης για τις επιχειρήσεις μας και για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται. Αν δεν μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι πολίτες μας, ποτέ δεν θα τις χρησιμοποιήσουν. Αν μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη σε αυτές τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, τότε θα τις χρησιμοποιήσουν. Και γι' αυτό ας το θυμόμαστε αυτό αυτή την περίπτωση Σούμαχερ που είναι ιδιαίτερα θλιβερή. Τα προσωπικά δεδομένα υγείας που εκλάπησαν σε σχέση με το άτομο αυτό, το Σούμαχερ. Ήταν σε έγγραφη, σε έντυπη μορφή αυτά τα στοιχεία, δεν είχαν ψηφιοποιηθεί και εκλάπησαν. Και θα ήθελα να πω σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το να κλέψει κανείς ένα είδος ε, πληροφοριών, να κλέψει πληροφορίες και να καταχραστεί πληροφοριών που είναι πολύ πιο εύκολο να κλαπούν από NDP μορφή από ότι να κλαπούν ε, ψηφιοποιημένα στοιχεία τα οποία έχουν προστατευτεί με ασφαλή τρόπο ψηφιακά. Ευχαριστώ. Τάγια Κάλλας, Άλντε από την ΕΜΚΟ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εστονικά. Στην αρχική σας παρέμβαση είπατε ότι μπορούμε να έχουμε κυβέρνηση, διακυβέρνηση χωρίς χαρτί. Ερώτηση, πόσο γρήγορα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μην χρησιμοποιεί πια χαρτί. Θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου δημιουργούμε τόνους χαρτούρας κάθε μέρα. Θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε πάρα πολύ χαρτί, πιστεύω, με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Για να υπάρξει πολυμορφία γλωσσική θα απαντήσω εσθονικά. Και πάλι πρέπει να πω για άλλη μια φορά. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε από μηδενικού σημείου. Όταν κάνουμε λοιπόν λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην χρησιμοποιεί πλέον έντυπο υλικό αλλά να ε, χρησιμοποιεί ηλεκτρονικής μορφής υλικά και ψηφιοποιημένα στοιχεία είναι πολλές φορές ε, ήδη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή έχουν προχωρήσει τα πράγματα αυτά. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές δυνατότητες να μειωθεί η χρήση έντυπων, ε, έντυπου υλικού, του χαρτιού, η χρήση εγγράφων σε έντυπη μορφή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για παράδειγμα, οι, λογαριασμοί ε, και η τιμολόγηση ηλεκτρονική έχουν διευκολύνει τη ζωή των πολιτών στην Δανία, στην Ισπανία, στην Φινλανδία και αλλού. Εμείς λοιπόν πρέπει να ξεκινήσουμε να χρησιμοποιούμε ηλεκτρονική τιμολόγηση και ηλεκτρονικούς λογαριασμούς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μια μέρα θα μπορέσει να επιτευχθεί αυτό και εδώ πιστεύω και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για παράδειγμα στην Επιτροπή Ήτρε είχα ε, θέσει το ερώτημα γιατί όταν για παράδειγμα αγοράζουμε ε, εισιτήρια αεροπλάνων να μην τα αγοράζουμε σε έντυπη μορφή, να τα αγοράζουμε ηλεκτρονικά. Γιατί θα ε, πρέπει να εκτυπώνονται τέτοιου είδους ηλεκτρονικά εισιτήρια σε σχέση με την διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για παράδειγμα. Και είμαι πεισμένος ότι αν μπορέσουμε να δώσουμε ένα θετικό παράδειγμα εμείς οι ίδιοι με ένα ρόλο πρωτοπόρων μπορούμε πολλά, να αλλάξουμε πολλά μπορούν να αλλάξουν και είμαι πεισμένος ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσουν να καταφέρουν να είναι υποδειγματικοί στο ρόλο τους ε, για αυτά τα οποία θα πρέπει να γίνουν και να μιμηθούν και άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Σπινέλη, κύριε Σπινέλη, από την ΚΟΕ, χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Για τη θεματολογία του ψηφιακού τομέα. Τι Μέρμαν Γιουρκοβά και εσείς θα είστε υπεύθυνοι. Τι μπορείτε να κάνετε στον τομέα αυτό, ώστε να υπάρχει μια χάρτα δικαιωμάτων του ίντερνετ ένα είδος ε, πολιτικού δηλαδή πλαισίου όπως αυτό που υιοθετήθηκε φέτος στη Βραζιλία. Δεν αρκεί νομίζω να δημιουργήσουμε μόνο μια αγορά. Δεν αρκεί να αποδείξουμε δηλαδή ότι είμαστε οι υπουργοί φιλελεύθεροι. Χρησιμεύουν, χρειάζονται μάλλον οι κανόνες, ιδιαίτερα στο ίντερνετ. Κανόνες που θα πρέπει να σέβονται ε, τις διαφορές, τη διαφορετικότητα, τα διάφορα δικαιώματα που απορρέουν από την ε, Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και αυτό το ρωτάω ακριβώς κατά πόσο θέλετε έτσι να δεσμευτείτε ώστε να δημιουργηθεί μια χάρτα δικαιωμάτων του ίντερνετ όπως ακριβώς στη Βραζιλία. Ευχαριστώ. Uh, yes, I think there... Ναι, πράγματι πρέπει να έχουμε μια χάρτα ιντερνετικών δικαιωμάτων στην Ευρώπη πολλές από τις αρχές που αναφέρατε βρίσκονται και σε κανισμούς, οδηγίες, Αυτές λοιπόν τις κύριες αρχές τις έχουμε στην Ένωση και νομίζω ότι όλοι βεβαίως θα πρέπει να προσθέσουμε εδώ και ένα κεφάλαιο που να αφορά τα Ιντερνετικά δικαιώματα. Αναφέρθηκαν προηγουμένως και στο θέμα της Ιντερνετικής ουδετερότητας. Εγώ είμαι περήφανος που θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που η Ιντερνετική ουδετερότητα θα ρυθμίζεται σε επίπεδο οδηγίας. Στην ομοθεσία μας δηλαδή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας. Τώρα για την πρόσβαση στο ίντερνετ. Νομίζω ότι είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα αυτό και πραγματικά θα πρέπει να περιγράφουμε αυτά τα δικαιώματα με τρόπο πιο λεπτομερή και συγκεκριμένο προς τους πολίτες μας. Οπότε η απάντησή μου είναι ναι και σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Mr. from the Greens από τους πράσινους Ίντρε. Right. Thank you, Mr. Anzik, for your smooth deliberation. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ώρες σας απαντήσεις. Έχω ένα μικρό πρόβλημα με τη γραπτή σας απάντηση. Ως πολίτης και ως πολιτικός ήμουν ανέκαθεν υπέρ του ευρωπαϊκού εγχειρήματος που βασίζεται στις ε, δημοκρατικές αξίες. Αυτό είπατε. Ω διαχειριστή ενό κομμουνιστικού κόμματο, ε, πραγματικά προωθούσατε τι δημοκρατικέ αξίε σε αυτά τα 10 χρόνια. Οπότε ε, υπάρχει μια ανακρίβεια εδώ στην απάντησή σα. Και τι εμπιστοσύνη ε, πιστεύετε ότι θα πρέπει να δείξουν τα μέλη εδώ του Κοινοβουλίου σε εσά όταν εσεί πλοφάρετε. Εγώ δεν ξέρω κατά πόσο έχετε καλέ προθήσει, αλλά λυπάμαι, λυπάμαι πραγματικά για την ασθένεια σα εδώ και σα εύχομαι καλή ανάρρωση. Ευχαριστώ. Το παρελθόν μου, κοιτάξτε, είναι διαφανές. Όλοι στον γνωρίζουν ότι ήμουν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Αλλά όλοι γνωρίζουν επίσης ότι ήμουν δήμαρχος δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Εστονίας κατά τη διάρκεια έξι ετών και επανεξελέγην. Όλοι γνωρίζουν επίσης την Εστονία ότι εγώ εξελέγην τέσσερις φορές βουλευτής. Όλες οι λεπτομέρειες είναι γνωστές για το παρελθόν μου. Οι πολίτες της χώρας μου στις πρόσφατες ευρωεκλογέ έδωσαν υψηλά ποσοστά στο κόμμα και σε μένα προσωπικά. Και το κόμμα μου δηλαδή και εμείς προσωπικά είχαμε ψηλή σταυροδοσία κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών στην Εστονία των περασμένων. Το παρελθόν μου λοιπόν είναι διαφανές και δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ευχαριστώ. Μπέγγεν e από το EFTD. Ευχαριστώ. Κύριε Παψήφιε Επίτροπε, η ψηφιακή αγορά αποτελεί, μάλλον περιλαμβάνει ένα πολλαπλασιαστή ανάπτυξη πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες. Αυτές οι επιχειρήσεις έχουν διπλό συντελεστή ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας. Μιλήσαμε προηγουμένως για την υψηλή ταχύτητα, για την πρόσβαση ιδιαίτερα στις περιοχές της υπαίθρου που δεν υπάρχει σύνδεση με το ίντερνετ το δυναμικό της διάδοσης των υψηλών συνδέσεων ε, σύνσταται και στο να πλησιάσουν περισσότεροι οι πολίτες στα κέντρα απόφασης ώστε να καταλήξουμε μια μέρα σε αυτή την άμεση δημοκρατία που εγώ ως εκπρόσωπος του κινήματος των πέντε αστέρων πιστεύω απόλυτα. Η πρόσβαση λοιπόν τις ευρωζωνικές ε, ταχύτητες πρέπει να διασφαλιστεί για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Τι προθέσετε να κάνετε γι' αυτό. Και επίσης δεν θεωρείτε ότι η αύξηση της νέας ψηφιακής αγοράς θα μπορούσε να συμβαδίσει με την χρήση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί και από τους πολίτες και από τη δημόσια διοίκηση. Ευχαριστώ. Thank you. Uh, Ευχαριστώ. Αναφερθήκαμε στο θέμα του ανοιχτού λογισμικού προηγουμένως. Η απάντηση είναι η ίδια. Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποστηρίξει την χρήση του ανοιχτού λογισμικού, θα δημιουργήσει θέσει εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πιο ευέλικτη η προσέγγιση από ότι το λογισμικό που χρειάζεται αδειοδότηση και από ό,τι καταλαβαίνω, αν δεν μιλάμε για ε, μαζική παραγωγή είναι και κάπως πιο φτηνό από ότι το αδειοδοτούμενο ε, λογισμικό. Πρέπει να βρούμε το σωστή ισορροπία μεταξύ του ανοιχτού λογισμικού και εκείνου που χρειάζεται αδειοδότηση. Τώρα, το χαμηλό κόστος αποστολής. Καμιά φορά το τέλος αποστολής είναι πολύ ψηλό. κυρίως για την πώληση στο εξωτερικό, στο Λονδίνο, Φερρυπίν. Με ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να αποκτήσει κανείς αγαθά εντός λεπτών. Σε κάποιες άλλες χώρες όμως, για συγκεκριμένα αγαθά και για τη χώρα που ξέρω καλύτερα, πρέπει να περιμένει κανείς και δύο εβδομάδες ακόμα. δυσανάλογο το κόστος αποστολής, πολύ ψηλό. Δεν πρέπει να δεχθούμε και να ανεχθούμε αυτή την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Ήπεθρο. Μιλήσαμε γι' αυτό ήδη. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το τελικό κομμάτι για να χρησιμοποιήσουμε σωστό δίκτυο και στην Ήπεθρο. Για το τελικό αυτό σκέλος που αναφέρατε. Ευχαριστώ. Είμαστε πέρα από το μισό του δρόμου. Πάμε στον τέταρτο γύρο ερωτήσεων από το ΕΛΚ, από τον κύριο Κοέλιο. Ευχαριστώ. Κύριε Χάνσιμ, κατά τα τελευταία τρία χρόνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πολύ μικρή πρόοδος επετέφθη όσον αφορά το, ε, τον αριθμό επίγουσας κλίσης 1-1-2 στην Ευρώπη. Είχαμε πρώτα την ε, πρώτη προσέγγιση. Δεύτερον, ε, ο Καλόν σε σχέση με διάφορα κράτη-μέλη αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια όσον αφορά την άμεση βοήθεια και η ενημέρωση, οι πληροφορίες που δίνουν στους πολίτες δεν επαρκούν και μόνο ένα μικρό ποσοστό των Ευρωπαίων πολιτών γνωρίζουν ποιο είναι, το, ποιος είναι ο αριθμός άμεσης βοήθειας, αριθμός κλήσης ε, άμεσης βοήθειας. Αν θέλουμε να μεριμνήσουμε υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών υπάρχει μεγάλο περιθώριο για να κάνουμε πολλά πράγματα και να σημειωθεί πρόοδος. λαμβάνοντα υπόψη τον ρόλο σας ως Επιτρόπου για τα ψηφιακά μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι οι επίγουσες ε, βοήθειες ε, και ο αριθμό κλήση 2 πανευρωπαϊκά θα είναι προτεραιότητα για εσά όσον αφορά την ψηφιοποιημένη ε, ευρωπαϊκή αγορά και αυτά θα έπρεπε να πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντάξει, σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Μάλιστα, απαντώ. Πιστεύω ότι το σύστημα ηλεκτρονικής κλήσης ως αριθμός άμεσης βοήθειας είναι πολύ σημαντική υπόθεση γιατί θα βοηθήσει να διασωθούν ανθρώπινες ζωές, να σωθούν ζωές. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, σας διασφαλίζω, ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτή η φιλοδοξία, αυτός ο στόχος. Αλλά για άλλη μια φορά και πάλι, το θέμα είναι θέμα εμπιστοσύνης και πάλι ή έλλειψης εμπιστοσύνης κιόλας κυρίως όσον αφορά τους πολίτες. Κάποιοι και φυσικά και κάποια θεσμικά όργανα δεν είναι βέβαιοι σήμερα ότι αυτά τα στοιχεία, δηλαδή για την ηλεκτρονική κλίση αυτοί οι αριθμοί δεν θα χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα για να εντοπιστούν άτομα καταχρηστικά. Πρέπει να προστατέψουμε λοιπόν την ιδιωτική ζωή και τη σφαίρα ιδιωτικότητας του καθενός. Πρέπει να προστατέψουμε όλα αυτά τα πολύ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και δεδομένα γενικότερα. Και αν θα είναι βέβαιοι οι πολίτες και θα υπάρχει ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και θα γνωρίζουν ότι θα προστατεύονται και οι ευρωβουλευτές επίσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάλι και όλα τα κράτη-μέλη ε, τότε θα υπερψηφίσουν λοιπόν και θα δράσουν υπέρ αυτής της ε, πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ. Νίκολα Ντάντι, from the S&D for ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπη, υπάρχουν τρεις βασικές προτάσεις από το οποίο το Κοινοβούλιο ήδη έχει τοποθετεί ξεκάθαρα. Νομοθετικό πακέτο για τις συνδέσεις στην Ήπειρο, διασύνδεση μάλλον της, Ήπειρο, της Ήπειρου, δημόσια διοίκηση και η ασφάλεια των δικτύων. Τρεις προτάσεις που μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην μείωση της απόστασης μεταξύ διοικήσεων, πολιτών και επιχειρήσεων, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, βοηθώντας την οικονομική ανάκαμψη και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες. Επ' αυτού είναι σημαντικό να επιτευχθούν φιλόδοξες συμφωνίες με το Συμβούλιο. Ποιες συγκεκριμένε προτάσεις και με ποιο πνεύμα προτείνετε να δράσετε ώστε να ευνοήσετε την ε, ταχεία εφαρμογή αυτών των προτάσεων μετά συγκεκριμένα σε σχέση με την οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων. Δεν θεωρείτε ότι μαζί με μια απαραίτητη συνεργασία σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να υπάρχει και μια μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία και εν της επιθυμητής ε, αναθεώρησης της δημόσιας διακυβέρνησης του κυβερνοχώρου. Ευχαριστώ. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την συνδεδεμένη Ήπειρο, για το πακέτο για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών και όπως υπογραμμίσαμε επανειλημμένα ήδη σήμερα, πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να δημιουργήσουμε μια ενιαία αγορά. Όλα τα στοιχεία λοιπόν του TCM είναι σημαντικά για την ενιαία αγορά κυρίως όταν μιλάμε για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την ουδετερότητα του δικτύου. Μετά. Α, το δεύτερο τμήμα της ερωτήσεως. Μπορείτε να το επαναλάβετε, παρακαλώ. Μπορείτε να επαναλάβετε. Τι δράσεις προτίθεστε να λάβετε, να δρομολογήσετε ούτω ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ Ευρώπης και του υπόλοιπου παγκοσμίου δικτύου. Και ίσως να υπάρχει και κάποια μορφή παγκόσμιας διακυβέρνησης ε, του διαδικτύου. Δεν το έπιασα αυτό το δεύτερο, το διεθνές κομμάτι της ερώτησης. Ξέρω ότι οι διαπραγματεύσεις για τον ασφαλή λιμένα ήταν περιπλοκότατες και δυσκολότατες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε 13 προτάσεις. Από τις 13 οι περισσότερες αφορούσαν θέματα επιχειρητικά. Αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα της εθνικής ασφάλειας και την εξαίρεση για εθνική ασφάλεια. Πρέπει να υπάρχει εξαίρεση για εθνική ασφάλεια. Εξαίρεση όμως. Όχι τακτικά. Και για όλα τα δεδομένα. Οι Αμερικανοί πρέπει τελικά να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους. Πρέπει να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης για τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει όμως να παραμείνει επιτάπητος και η πιθανότητα αναστολής των διαπραγματεύσεων. Επόμενη δική μου ερώτηση, λέει Πρόεδρος. Υποσχεθήκατε σε κάποιο συνάδελφο ότι θα είναι online η ακροασή σας. Αλλά πρέπει να σας αξιολογήσουμε σε αυτά που λέτε απόψε αλλά επειδή πιστεύω στην ψηφιακή επαφή με το κοινό, ρώτησα κάποιους κατά τη διάρκεια, βάθησα ερωτήσεις ανθρώπους από το Twitter. Μας θέσανε ερωτήσεις για τη περιαγωγή, για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και για το πόσο πρέπει να προσαρμόζεται με μελλοντικέ εξελίξεις η νομοθεσία. Λοιπόν, από, οργανώσει οργανω... από οργανώσεις ε, εταιριών για την νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων έρχονται ερωτήσεις στο Twitter και πώς θα πετύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά, ε, κυρίως όσον αφορά ανησυχίες που ακούγονται από τις μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή πώς μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία καταναλωτών για να μπορούν να προωθήσουν το ηλεκτρονικό εμπόριο από τη μια, αλλά να προστατεύσουν και τα συμφέροντα του καταναλωτού από την άλλη. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. η προστασία δεδομένων, όπως ήδη προανέφερα. δεν αναφέρεται σε σχέση με τις υπηρεσίες και οργανισμούς προστασίας δεδομένων. Η πραγματική προστασία δεδομένων είναι και υποστηρίζει όλες τις επιχειρήσεις, άσχετα από το μέγεθός τους, μεγάλες ή μικρές επίσης επιχειρήσεις που προστατεύονται από την προστασία δεδομένων. Προστασία δεδομένων. Προστασία της ιδιωτικής ζωής και σφαίρας του κάθε πολίτη. Η εμπιστοσύνη είναι τα θεμέλια των λύσεων στα ψηφιακά και στα ηλεκτρονικά και των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται. Χωρίς προστασία δεδομένων δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να πετύχει και να έχει να ε, ηγείται μιας επιτυχούς ε, εταιρείας, μιας επιτυχούς επιχείρησης. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία πραγμάτων μεταξύ των συμφερόντων των πολιτών μας που πρέπει να προστατευτούν και των συμφερόντων των επιχειρήσεων. Και πάλι δεν πρέπει να ξεκινήσουμε από μηδενικού σημείου. Είναι μια ενρευστό σε εξέλιξη ευρισκόμενη διαδικασία και μετεξελίσσεται και νομίζω ότι κινούμεθα με ταχύς ρυθμούς και ταχαίως προχωρούμε σε σχέση με αυτά τα θέματα. Φυσικά όλοι θα επιθυμούσαμε και θα θέλαμε να υπάρχουν ε, διατάξεις και κανονισμοί ήδη έτοιμοι προτού ε, υπάρξουν κάποιες πραγματικές τεχνικές δυνατότητες δράσης. Όμως από την άλλη πλευρά δεν είναι εφικτά τα πάντα, δεν είναι όλα δυνατά να γίνουν. Θα κάνω λοιπόν πραγματικά ό,τι μπορώ, ό,τι περνάει από το χέρι μου, να βρω τη σωστή ισορροπία που θα εξεύρω και θα διασφαλίσω μεταξύ προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων και προστασίας συμφερόντων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ. Morgan Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Άνσιπ. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο καινοτόμα, πιο ανταγωνιστική και πιο ανοιχτή και πιο διαφανής Χρειάζεται λειτουργικότητα και ανοιχτέ προδιαγραφέ. Είναι κρισίμου σημασία για να αναπτυχθεί η Ευρώπη και να γίνει ανταγωνιστική και ανοιχτή στην αγορά. Θα στηρίζατε να αντιμετωπιστεί η διαλειτουργικότητα και η χρήση ανοιχτών εγγράφων πιο συστηματικά και από όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και οι ανοιχτέ αυτέ προδιαγραφέ τι ρόλο μπορούν να παίξουν Πιστεύετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουν ε, ανοιχτές υποδομές και προδιαγραφές σαν κοινοτικά όργανα. Γενικότερα, τι θα κάνετε να υποστηρίξετε και να προωθήσετε τις ευρωπαϊκές εταιρείες και μια ευρωπαϊκή πολιτική για προστασία των δεδομένων και προστασία της ιδιωτικής ζωής στο συζητούμενο πλαίσιο. Απάντηση, ευχαριστώ. Διαλειτουργικότητα σε πολλές περιπτώσεις είναι λέξη κλειδί. Υπάρχουν σε κράτη-μέλη διάφορες λύσεις που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο αλλά δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σε κάποιες άλλες φορές Θα ήθελα ξανά να μιλήσω για τη δική μου χώρα. Κάθε χρόνο 20.000 Εστονοί εργάζονται σε γειτονική χώρα και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να φέρουν κάποια έγγραφα από το ληξιαρχείο μας και να το πάνε στη γειτονική χώρα. Λόγω ελλείψεως διαλειτουργικότητας. Αυτό είναι αδύνατον. Σημαίνει ότι αυτοί που εργάζονται στη γειτονική χώρα και πολύ ανεπτυγμένη χώρα είναι αυτή. Αναπτυγμένη όσον αφορά τα ψηφιακά, την ψηφιακή τεχνολογία. Φιλανδία. Κάθε χρόνο 20.000 άνθρωποι που εργάζονται στη Φιλανδία πρέπει να αγοράσουν εισιτήρια για το ferry boat, για το αεροπλάνο, να πάνε στην Εστονία και στην πρεσβεία μας στη Φιλανδία μπορούν να το το θέμα τους. Τέλος πάντων, έρχονται στην Εστονία, περιμένουν στην ουρά για να πάρουν τα αναγκαία έντυπα με υπογραφές, με σφραγίδε. και μετά ξανά στο οχηματογωγό του, πάνε στη Φιλανδία και στη Φιλανδία οι δημόσιοι υπάλληλοι περνάνε τα στοιχεία προσεκτικά στους υπολογιστές τους και ξανά γίνεται ψηφιακή πληροφορία. τον 21ο αιώνα γιατί να είναι στα πράγματα, κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Και δεν πρέπει να είναι έτσι, θα πρέπει να προωθήσουμε τη διαλειτουργικότητα. Ευχαριστώ. Κονίλια Έρνστ, της ΓΚΟΕ, Επιτροπή Βιομηχανίας. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και πάλι να επανέλθω στην προστασία δεδομένων, προσωπικών δεδομένων και για την αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μεταρρύθμιση της προστασίας ε, προσωπικών δεδομένων ώστε συμφωνίες και συμβάσεις που αφορούν προσωπικά δεδομένα να καλύπτουν αυτά τα θέματα. Και το Κοινοβούλιο έχει λάβει μια τέτοια απόφαση ε, όπου συμπεριλαμβάνεται ότι όποιος επεξεργάζεται ευρωπαϊκά δεδομένα θα πρέπει να σέβεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αυτά όλα αντιφάσκουν, βρίσκονται σε αντίφαση με πολλές συμφωνίες που υπάρχουν και βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση. Πρώτη ερώτηση. Πιστεύετε ότι οι συνθήκες και συμφωνίες όπως το Safe Harbor, ο ασφαλής λιμένας, που υπονομεύουν το επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν δίνουν καθόλου εχέγγυα για την προστασία τους. Ότι θα πρέπει τέτοιου είδους συνθήκες και συμφωνίες ε, να αλλάξουν ή να αναδιαρθρωθούν, να αναδομηθούν. Και για την συμφωνία TTIP, για την ε, συμφωνία ελευθέρου εμπορίου και επενδύσεων με τη ΣΥΠΑ, πρέπει να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο επίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αναφέρθηκα σήμερα στο safe harbor στο ασφαλή λιμένα. Όμως αυτό δεν είναι πια ασφαλή σήμερα. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε στην Ευρώπη ότι αυτός ο ασφαλής λιμένας δεν είναι για τόσο ασφαλή σήμερα. Οπότε θα ε, πρέπει να τον κάνουμε πραγματικά ασφαλή το λιμένα τον ασφαλή. Αλλά για τον κάνουμε ασφαλή το λιμένα τον ασφαλή επιχειρήσεις και οι πολίτες θα πρέπει να ενδιαφερθούν σε αυτό. Θα πρέπει πραγματικά να γίνουν αλλαγές στον υπάρχοντα ασφαλή λιμένα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέβαλε 13 προτάσεις και η πλειοψηφία τους ε, έτυχε θετικής απάντησης. Οπότε ακόμα και αυτές οι προτάσεις που έλαβαν θετικές, προτάσεις, θετικές ε, απαντήσεις θα μπορούσαν να μας κάνουν το λιμένα τον ασφαλή ασφαλέστερο. αλλά όχι φαίνεται, δεν φαίνεται όμως να είναι επαρκώς ασφαλής γιατί οι πολίτες μας ανησυχούν για αυτές τις εξαιρέσεις εθνικής ασφάλειας ας πούμε δεν ξέρουν πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι εξαιρέσεις για λόγους εθνικής ασφάλειας. Τώρα περιμένουμε να γίνουν κάποια έτσι ουσιώδη βήματα από την πλευρά των Αμερικανών. Εάν εμείς δεν δεν λάβουμε σαφείς απαντήσεις για το πώς αυτές οι εξαιρέσεις ε, εθνικής ασφαλείας θα χρησιμοποιηθούν, τότε βεβαίως η διακοπή ως ε, επιλογή θα πρέπει να παραμείνει έτσι υπαρκτή σαν ενδεχόμενο. Λίμπε, πράσινη, Βέρκ. Αγαπητέ κύριε σας ευχαριστώ πολύ για τη στεναρή σας τοποθέτηση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε την τεράστια πλειοψηφία του σώματος που σας υποστηρίζει για να προχωρήσετε. Έχουμε υπεψηφίσει το πακέτο προστασίας δεδομένων με υψηλές προδιαγραφές. Πρώτη ερώτηση, πώς θα μπορέσετε να αποφύγετε ότι το Συμβούλιο των Υπουργών θα διαφωνήσει και θα βρεθεί πολύ μακριά, θα παρεκκλίνει σημαντικά από την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς εμείς έχουμε κάποιες ε, κόκκινες διαχωριστικές γραμμές για τις θέσεις μας και θέλουμε να είναι σεβαστές ε, και για το open source, ε, τις ανοιχτές πηγές. Πώς θα διασφαλίσετε ότι προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται στις ευρωπαϊκές αγορές δεν θα ανοίξουν πόρτα και παράθυρο, για παράδειγμα, να υπονομευθούν αυτές οι προδιαγραφές μας. Η μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υποστηρίζει τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων. Όπως βλέπω τα πράγματα, τα καλά μαντάτα είναι ότι όλο και περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν την προστασία των δεδομένων και τα σχετικά πλαίσια. Υποσχέθηκα να κάνω ό,τι μπορώ ούτως ώστε να εξεύρω καλές λύσεις για τους πολίτες μας. Είμαι βέβαιος ότι οι πρώην συνάδελφοί μου θα ήθελαν να, δουν να πραγματοποιείται η ψηφιακή ενιαγόρα. αγορά. Αλλά είναι ανέφικτο αν δεν υπάρχει μεγάλη ασφάλεια για την προστασία των δεδομένων. Η προστασία των δεδομένων είναι προϋπόθεση για την ενιαία ψηφιακή αγορά. Το λογισμικό ανοιχτής πηγής σαν τη Wikipedia είναι. Όλοι μπορούν να πάνε στη Wikipedia, να τη χρησιμοποιήσουν, να τη συμπληρώσουν, να αναπτύξουν. Και αν ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιήσει και να αναπτύξει το λογισμικό, όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, είναι κάπως πιο ευάλωτο το λογισμικό. Με το λογισμικό που χρειάζεται άδεια όμως είναι πιο περίπλοκο να βρει κανείς τις χερκόπορτες και να κάνει hacking. Είναι θέμα εμπιστοσύνη. Πρέπει να δημιουργήσουμε πραγματική εμπιστοσύνη εδώ στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Dario Tamburano from the EFDD, from the Industry Committee. Tamburano EFDD, Επιτροπή Μηχανίας. Γεια σας, Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τον συνάδελφό μου. Κύριε Πίτροπε, Εσεί είστε υπεύθυνοι της ενιαίας ψηφιακής αγορά. Εμεί θα θέλαμε να θίξουμε μια συγκεκριμένη πτυχή αυτή τη αγορά, δηλαδή το ίντερνετ. Το ίντερνετ δεν είναι μόνο ένας χώρος όπου γίνονται αγοραπολισίε αγαθών, υπηρεσιών ή ψυχαγωγίε. Κατά την άποψή μα. το ίντερνετ σαν το νερό είναι κοινό αγαθό αγαθό δηλαδή κοινή ωφέλεια. Το ίντερνετ είναι απαραίτητο όταν ένα πολίτη θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τι ε, δημόσιε αρχέ, όταν θα πρέπει να έχει πρόσβαση ε, στην επικαιρότητα, στη γνώση, στον πολιτισμό. Είναι ένα τρόπο δηλαδή για να μείνουμε έτσι κοντά όταν είμαστε μακριά. Ρωτάμε λοιπόν, δεσμεύεστε για αυτέ τι πτυχέ να δηλώσετε ότι αποτελούν ένα κοινό αγαθό εκτό δηλαδή νόμων τη αγορά. Thank you. Διαδίκτυο πρέπει να είναι πάντα ανοιχτό και όλοι να μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό χωρίς αποκλεισμούς. Και φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατέψουμε την πολιτισμική μας ποικιλότητα, ποικιλομορφία και νομίζω ότι επιτυχώς ε, το προσπαθούμε και το πετυχαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό. Το ερώτημα σας τώρα ήταν και αφορούσε επίσης και την διακυβέρνηση στο διαδίκτυο. Είμαι υπέρμαχος του πολλαπλού προτύπου των εμπλεκόμενων δηλαδή που θα μπορούν να συνεισφέρουν στην διακυβέρνηση του διαδικτύου. Πολλές ε, χώρες και πολλές ε, προσπάθειες γίνονται για να αλλάξει αυτό το πρότυπο σε ένα διακυβερνητικής μορφής πρότυπο. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε την αλλαγή αυτού του πλαισίου όπου όλοι θα μπορούν να συμμετέχουν, ακόμα και μη κυβερνητικές οργανώσεις, στην διακυβέρνηση, στην διαχείριση. Η αλλαγή στο διακυβερνητικό πλαίσιο θα μπορούσε να είναι θετική για το διαδίκτυο. Όμως θα πρέπει να αλλάξει το σημερινό πρότυπο, να γίνουν κάποιες αλλαγές για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Σήμερα πιστεύω σε κάποιες χώρες δεν εμπλέκονται τόσο πολύ και δεν συμμετέχουν τόσο πολύ στη διακυβέρνηση και διαχείριση του διαδικτύου. Και επίσης και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να μεγεθυνθεί, να αυξηθεί. Ευχαριστώ. last 15 questions. 15 ε, ερωτήσεις. Στέφανες, Ινκο, Ελκ. Σας ευχαριστώ. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, με μεγάλη ικανοποίηση άκουσα στις αρχικές σας εισαγωγικές παρατηρήσεις το θέμα της ηλεκτρονικής υπογραφής. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι η ηλεκτρονική υπογραφή είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο για να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτών των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών. Γι' αυτό η ερώτησή μου είναι ποια συγκεκριμένα βήματα και διαβήματα θα κάνετε ώστε να εφαρμοστεί και να προαχθεί η ηλεκτρονική υπογραφή, ώστε να απλουστευτούν οι διαδικασίες που ισχύουν. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Και πάλι φέροντας ένα παράδειγμα σε σχέση με την χώρα μου. Δώσαμε στους πολίτες μας εμείς στην Εσθονία υψηλού επίπεδου ε, προστατευόμενες ε, ψηφιακές ταυτότητες και εφαρμόσαμε την εφάπαξ αρχή νομικά και μάλιστα το 2007 το ξεκινήσαμε αυτό στην ε, Εσθονία. Και σήμερα όλοι πλέον χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπογραφές στην Εστονία. Ήδη οι Εστονοί πολίτες έδωσαν, συνέλεξαν από το 2002 175 εκατομμύρια διαδικτυακά ηλεκτρονικές ε, υπογραφές ε, ενώ είμαστε ε, από πλευράς πληθυσμού στο επίπεδο των τριών περίπου εκατομμυρίων και πρέπει να δούμε ότι αυτό έχει συνεισφέρει το να εξοικονομείται μία εβδομάδα εργασίας ανά Είναι πολύ μεγάλη αυτή η πρόοδος και για τις αμυντικές μας δαπάνες. Μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη εξοικονόμηση και καλή καλύπτονται μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών και μάλιστα έχει προχωρήσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με αυτόν τον κανονισμό λοιπόν, οι ηλεκτρονικές ταυτότητες πρέπει αμοιβαία να αναγνωρίζονται ε, με βάση συγκεκριμένες προδιαγραφές, να είναι αμοιβαία ε, αποδεκτές. Και αυτό θα είναι και είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός να οδηγηθούμε στο ότι αυτή η ηλεκτρονική υπογραφή να μπορεί να χρησιμοποιείται πανευρωπαϊκά σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επιπρέφη Επίτροπε, όπως επανειλημμένως υπογράμμισε το Κοινοβούλιο, η ολοκλήρωση της νέας ψυχική αγορά θα οδηγήσει σε αύξηση απασχόληση και τη ανάκαμψη. Όμω αυτή η αγορά δεν αποτελεί μόνο ευκαιρία για του πολίτε και τι επιχειρήσει, πρέπει να αποτελεί μια ευκαιρία για τι δημόσιε αρχέ και σε ευρωπαϊκό και σε ε, εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Ο εξυγχρονισμό των ευρωπαϊκών δημοσίων αρχών και η ανάπτυξη δημοσίων υπηρεσιών online που θα είναι αποτελεσματικέ είναι απαραίτητε για να ανταποκριθούμε σε κοινέ ανάγκε των πολιτών και των επιχειρήσεων. Άκουσα, είπατε στην αρχή την βούλησή σας να ενθαρρύνετε ακριβώς την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική διοίκηση. Ποια είναι λοιπόν τα μέτρα που θα λάβετε για να διασφαλίσετε, να διασφαλίσετε ότι η ψηφιοποίηση και ο εξυγχωρισμός της δημόσιας διοίκησης πραγματικά θα υλοποιηθούν για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ιδιαίτερα τα εννέα σημεία επαφή που προβλέπουν οι οδηγίες για τις υπηρεσίες και την αμοιβαία αναγνώριση των ε, επαγγελματικών προσόντων, ώστε να επιτρέψουμε την κυκλοφορία των επιχειρήσεων αυτών των υπηρεσιών, διασφαλίζοντα την ποιότητά του και συγκεκριμένα προστατεύοντα και του καταναλωτέ, Ποια μέτρα λοιπόν συγκεκριμένα προτίθεται να αναλάβετε προ την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ. Σήμερα αναφερθήκαμε σε κάποια παραδείγματα και τις δυνατότητες που παρέχουν. Θα δώσουμε ένα παράδειγμα λοιπόν βεβαίω στους πολίτες μας και στις χώρες μέλη για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το e-governance. Αυτές λοιπόν οι λύσεις που παρέχονται μέσω ίντερνετ, δημόσιες υπηρεσίες ας πούμε, θα πρέπει να είναι χρήσιμες στους πολίτες μας. Αν λοιπόν ο κόσμος τα, βρέπει θετικά θα αρχίσει να τα χρησιμοποιεί. Και πάλι να αφαιρθώ στο παράδειγμα της Εστονίας. Όταν εφαρμόσαμε το ηλεκτρικό φορολογικό σύστημα στην Εστονία, τότε τον πρώτο χρόνο ήταν έτσι πολύ δημοφιλές το σύστημα αυτό στους πολίτες μας. πριν από αυτό το σύστημα ο κόσμος πήγαινε τις δηλώσεις του στις ΔΟΗ. Δεν είχαν εμπιστοσύνη στις ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ήθελα να είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει κανένα λάθος στις φορολογικές τους δηλώσεις. Τώρα, τώρα, ηλεκτρονικά συμπληρώνονται οι φορολογικές δηλώσεις στο ίντερνετ. Πανεύκολο είναι. Μισό λεπτό χρειάζεστε για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αυτά τα δεδομένα. Σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν γίνεται. Και μπορεί να είστε απόλυτα βεβαίως ότι δεν κάνατε κανένα λάθος και ότι κανείς θα σας βάλει πρόστιμο ή θα σας βάλει στη φυλακή. για τους τίμιους φορολογόμενους και τους έντιμους φορολογόμενους δουλεύει μια χαρά αυτό το σύστημα. 96% φέτος των δηλώσεων υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω αυτού του συστήματος των κοινωνικών δηλώσεων. Οπότε αυτές οι υπηρεσίες λοιπόν θα πρέπει να είναι ε, ωφέλιμες για όλους τους πολίτες, για όλους τους πελάτες μας. Τζαζανόσκι, Επιτροπή Βιομηχανία, CCR. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι στην ψηφιακή εσωτερική αγορά θέλετε να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα. Στο προηγούμενο κοινοβούλιο επιμακρό συζητήσαμε για την διασύνδεση των ευρωπαϊκών χωρών Connecting, Connecting Europe Facility και μετά περικόπηκαν τα κονδύλια. Δηλαδή δύο προγράμματα δεν μπόρεσαν να υποστηριχθούν και να ολοκληρωθούν. Ήταν προγράμματα για την υποστήριξη, για παράδειγμα, ταχαίως ευρυζωνικού δικτύου που θα θέλαμε ιδιαίτερα σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας ε, της Ασίας να προσεγγίσουμε τα δικά τους επίπεδα και να προοδεύσουμε. Το δεύτερο πρόγραμμα ήταν η υποστήριξη του ευρυζωνικού δικτύου στην Ήπεθρο, όχι στα μεγαλαστικά κέντρα αλλά εκεί όπου η αγορά δεν δίνει την δυνατότητα να υπάρξει ε, ιδιαίτερη υποστήριξη. Πώς συγκεκριμένα αυτά τα προγράμματα στο μέλλον θα τα υποστηρίξετε και θα τα ενισχύσετε ώστε να μην απολεστούν. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν έχουμε αρκετούς πόρους να καλύψουμε όλη την Ευρώπη με πάρα πολύ ταχείες ευρυζωνικές υπηρεσίες με το Connecting Europe Facility. Έχουμε άλλες πηγές όμως. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στον ορίζοντα 2020 όχι απλώς για την ευρυζωνική αλλά για το ψηφιακό τομέα υπάρχουν ε, σημαντικά ποσά τα ευρωπαϊκά διευθυντικά ταμεία διαθέτουν πόρους για τον ευρυζωνικό τομέα. Αν θέλουμε όμως να καλύψουμε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 100 MB ανά δευτερόλεπτο ευρυζωνικής υπηρεσίας τότε χρειαζόμαστε τουλάχιστον 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστιο ποσό. Αλλά αν δούμε τι κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δεν χρησιμοποιούν τα χρήματα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τα δίκτυα της ευρυζωνικής. Χρησιμοποιούν δημοτικά χρήματα, όχι της ομοσπονδιακής κυβερνήσεως. Σε άλλες χώρες, στην Αυστραλία Φερρυπίν, στην Ιαπωνία, στην Νότια Κόρια... χρησιμοποιούνται οι πόροι, οι δημόσιοι, για τη δημιουργία των ε, ευρυζωνικών δικτύων. Από τα χρήματα των ε, φορολογουμένων χρηματοδοτούνται. Ο υποψήφιος αντιπρόεδρος, ο κ. Κατάινεν, πρέπει να ετοιμάσει μια μεγάλη δέσμη μέτρων επενδυτικών. 300 δισεκατομμύρια ευρώ για ψηφιακούς σκοπούς. Ελπίζω ότι θα πάρουμε περίπου 35 από το πακέτο. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Ήδη μοιραζόμαστε τα χρήματα. Με μόχλευση μπορούμε να αυξήσουμε το ποσό και να φτάσουμε 130 δις. Α, τελείωσε ο χρόνος μου, λυπάμαι. Θα μοχλεύσουμε λίγο την ερώτηση, λέει Πρόεδρος. Επόμενος, παρακαλώ. Για την ΑΛΔΕ, Επιτροπή Βιομηχανίας. Η κυρία Νόβενχάζεν, ακούσαμε τις απαντήσεις σας και φαίνεται ότι είναι όφελος το ότι κατάγεστε από μια χώρα που είναι στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής ε, οικονομίας από την Εστονία είναι από ε, η Εστονία. Λοιπόν, το πρόβλημα του πληθυσμού είναι η γύρανση. Ποτέ πριν στην ιστορία δεν είχαμε τόσο πολλούς ηλικιωμένους. Αυτό συνεπάγεται πολλές προκλήσεις νέες για την ε, περίθαλψη της υγείας. Σε αυτό το τομέα τι θα κάνετε, στηρίζετε το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγολόγησης που χρησιμοποιείται σε κάποια κράτη-μέλη και πώς θα μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο ε, διασυνοριακά. Σας ευχαριστώ. Φυσικά υποστηρίζω την πρόταση και την προσέγγιση της, των λύσεων ηλεκτρονικού χαρακτήρα. Στην Σουηδία, για παράδειγμα, όταν υλοποίησαν, όταν εφήρμοσαν αυτές τις ε, συνταγές ηλεκτρονικά, ήταν πολύ δημοφιλής ευθύς εξ αρχής. Το ίδιο συνέβη και στην Ελλάδα. Όταν εφαρμόστηκε η ίδια μορφή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ε, υπήρξε αύξηση του αριθμού των ασθενών που χρησιμοποιούσαν τις ηλεκτρονικές ε, συνταγές και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Στη χώρα που γνωρίζω καλύτερα, την Εστονία, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ήταν ένα αρκετά περίπλοκο σύνθετο ζήτημα πληρώναμε, η κυβέρνηση πλήρωνε για την λύση των ηλεκτρονικών συνταγών συνταγογράφησης λιγότερο από ένα εκατομμύριο, όχι ένα δισεκατομμύριο, λιγότερο από ένα εκατομμύριο ευρώ. Και φυσικά αντιμετωπίσαμε και τεχνικού χαρακτήρα προβλήματα κατά την, φάση εφαρμογής και υλοποίησης της ε, ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στην Εστονία. Όμως σήμερα από την άλλη πλευρά όλοι οι πολίτες μας, όλοι οι Εστονοί είναι πραγματικά ικανοποιημένοι με αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης. Σε κάποιες περιπτώσεις για παράδειγμα δεν πρέπει να, έχει, να προστρέχει κανείς τον ε, οικογενειακό του γιατρό. Με ένα τηλεφώνημα απλό και χρησιμοποιώντας την ταυτότητά του μπορεί κανείς να έχει από κάθε γιατρό τη δυνατότητα συνταγογράψης αυτών των φαρμάκων. Λειτουργεί πραγματικά και διευκολύνει την ζωή των πολιτών μας πραγματικά και την καθιστά πολύ πιο εύκολη. Αναφέρατε επίσης και το θέμα της ε, γύρανσης του πληθυσμού. Υπάρχει ένας τεράστιος τομέας Δηλαδή η αργυρή οικονομία, η ασημένια οικονομία, όπου τα ψηφιακά μπορούν να έχουν θαυματουργά αποτελέσματα. Um, Ελπίζω να το έχουμε το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εύα Πανόβα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υποψήφιε Αντιπρόεδρε εδώ μπροστά σας, δεξιά, εδώ είμαι. Όπως ακούσαμε και όπως γνωρίζουμε, η χώρα σας, η Εστονία, είναι ιστορία επιτυχίας όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις κοινοβουλευτικές εκλογές. Θες στη χώρα μου, τη Βουλγαρία, ήμασταν μάρτυρες πάρα πολύ χαμηλής προσέλευσης των ψηφοφόρων. Για να αλλάξει η τάση προφανώς δεν χρειάζεται μόνο να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της πολιτικής αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζουμε τη συμμετοχή στην συμμετοχική δημοκρατία. Σαν βουλευτής εγώ θέλω να ολοκληρωθεί η ψηφιακή αγορά και πιστεύω ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί να πετύχει διαφάνεια, έλεγχο και απόδοση. Συμφωνείτε ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα ψηφοφορίας στα κράτη-μέλη θα προωθήσουν τη συμμετοχή του λαού στην πολιτική διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να στηρίξει και να δώσει κατευθύνσεις για την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων σε κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται κάτι τέτοιο. Και τι συγκεκριμένε δράσεις θα αναλάβετε τόσο ώστε να υποστηρίξετε ε, την εξάπλωση αυτών των, ε, της ηλεκτρονικής Σας ευχαριστώ πολύ. Συστήματα για τη συμμετοχή στις εκλογές ε, και την έκφραση ψήφου ηλεκτρονικά από πλευράς των ψηφοφόρων ως ε, υποψήφιος αντιπρόεδρος δεν επιθυμώ να πω ότι σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά δυνατότητες ψήφισης ε, και έκφρασης ψήφου των πολιτών. Είναι θέμα των κρατών μελών να αποφασίσουν και πώς θα ρυθμίσουν αυτόν τον τομέα. Όμως, εγώ είμαι υπέρ των ηλεκτρονικών εκλογών, ατομικά. Για πρώτη φορά στην χώρα από την οποία προέρχομαι και γνωρίζω καλύτερα το 2005 έγινε αυτό. Παρήχαμε σε όλη την Εσθονία δυνατότητες οι πολίτες ηλεκτρονικά να μπορούν να ψηφίσουν κατά τη διάρκεια των δημοτικών εκλογών. Και μόνο 10.000 πολίτες τότε ψήφισαν ηλεκτρονικά. Αλλά όπως επανέλαβα πολλάκις μέχρι σήμερα είναι θέμα εμπιστοσύνης, πλαισίου εμπιστοσύνης. Αν μπορούν να ε, εμπιστευθούν ότι τα χρήματα τα οποία διακινούν στο διαδίκτυο ότι είναι ασφαλή, ε, τότε και την ψήφο τους μπορούν να εμπιστευθούν ότι μπορούν να την εκφράσουν ηλεκτρονικά στο διαδίκτυο. Και κατά, τα τελευταία, κατά τις τελευταίες ε, εκλογές για το Ευρωκοινοβούλιο, είχαμε περίπου ένα τρίτο όλων των ψήφων που συνελέγησαν ηλεκτρονικά, με ηλεκτρονικό σύστημα από πλευρά των πολιτών που συμμετείχαν ηλεκτρονικά στην ψηφοφορία. Είμαι βέβαιος ότι σίγουρα πρέπει να παράσχουμε περισσότερες δυνατότητες να μπορούν να συμμετάσχουν στη δημόσια ζωή οι πολίτες ε, μέσω διαδικτύου. Και εκείνοι, για παράδειγμα στη χώρα από την οποία προέρχομαι και γνωρίζω καλύτερα την Εστονία, δεν είναι οι νέοι και οι νεότεροι, είναι οι πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι στη χώρα μου που έχουν εξοικειωθεί και με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε υποψήφι Επιτροπέ. Παρουσιάσατε μια στρατηγική για την πρόοδο της ενιαίας ψηφιακής αγορά και είναι μοναδική πραγματικά ευκαιρία που σα παρέχει η θέση σας ω αντιπρόσωπο για να συνεργαστείτε με του υπόλοιπους ε, επιτρόπους ώστε να εργαστείτε σε συγκεκριμένου τομεί. Έχω λοιπόν και εγώ συγκεκριμένα ερωτήματα για αυτό το θέμα. Μόνο το 14% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, εμπορεύονται στο ίντερνετ. Αυτό δεν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Προβλήματα όπω α πούμε θέματα διαχείριση του εμπορίου από τι μικρομεσαίε και δεύτερον χρηματοδότηση για τον εξοπλισμό των υποδομών του, ώστε να έχουν πρόσβαση στι ηλεκτρονικέ αγορέ. Υπό την άποψη αυτή θεωρώ ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν περιφερειακά κονδύλια ή κονδύλια από το Προκαταμείο Συνοχή για τι μικρομεσαίε. Δεύτερον, με τι νέε ευκαιρίε υπάρχουν και νέα προβλήματα, νέε πραγματικότητε. Η ισότητα των ευκαιριών στον ηλεκτρονικό τομέα Πώς εσείς προτίθεστε να μειώσετε αυτή την ανισότητα μεταξύ των γενεών, δηλαδή ύπεθρος, αστικές περιοχές, ώστε ακριβώς το, ο ψηφιακό ο κόσμο να μην αποτελέσει άλλο ένα παράγοντα έλλειψη ισότητα στην Ευρώπη. Μετά για τη δημιουργία τη ενιαίας ψηφιακή αγορά, αυτή η αγορά θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική και θα πρέπει να υπάρχουν παρόμοια κόστη στην Ευρώπη. Πώ θα οδηγήσετε λοιπόν του μεγάλου οργανισμού να μειώσουν, να μειώσουν τα κόστη, να υπάρχει ανταγωνιστικότητα σε αυτό το μέσο στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πραγματικά συμβαίνει ότι μόνο 14% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων πολλούν και συναλλάσσονται διαδικτυακά, ηλεκτρονικά. Και κυρίως τι συμβαίνει. Αυτό το ποσοστό είναι τόσο χαμηλό επειδή έχουμε μια κατακαιρματισμένη αγορά. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο να πωλήσει κανείς διασυνοριακά τα εμπορεύματά του και να συναλλάσσεται διασυνοριακά με μια τόσο κατακαιρματισμένη αγορά. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το γεγονός οπωσδήποτε. Και φυσικά υπάρχει και απουσία εκπαιδευμένων και καταρτισμένων σε δεξιότητες ηλεκτρονικές των πολιτών μας και πρέπει πολύ σοβαρά να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα ώστε να κινητοποιηθούμε και να μπορέσουμε να καταρτήσουμε περισσότερους πολίτες στα ηλεκτρονικά. Και όπως είπα στον ενακτήριο λόγο μου, το 2020 900.000 θέσεις θα απαιτούνται σε αυτόν τον τομέα, θέσεις εργασίας και θα πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον υπιαγωγείο ή από τους βρεφικούς σταθμούς από πολύ πρώιμη ηλικία ώστε να μπορούν οι μαθητές στα σχολεία να εξοικειωθούν και να καταρτιστούν και να εκπαιδευτούν και ευρύτερα ακόμα πρέπει να στρέψουμε μεγαλύτερη προσοχή στην δημιουργικότητα και στην εφάνταστη δράση των μαθητών στα σχολεία πολύ περισσότερο από ό,τι κατά τα τελευταία χρόνια, 20 χρόνια, διότι σήμερα πλέον δεν υπάρχουν σαφείς διαχωριστικές γραμμές στις επιστήμες, μεταξύ επιστημών και τεχνών για παράδειγμα, καλών τεχνών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια για, από πλευράς περιφε, Ταμείου Περιφερικής Ανάπτυξης, από το Κοινωνικό Ταμείο επίσης, για να δημιουργήσουμε δυνατότητες υποστήριξης και ενδυνάμωσης του ψηφιακού ηλεκτρονικού τομέα. Και κάνουμε χρήση αυτών των κονδυλίων ήδη σήμερα. Η διαβίου μάθηση και εκπαίδευση επίσης, lifelong learning, είναι κάτι που πρέπει πολύ σοβαρά να το δούμε και να το προσεγγίσουμε. Και αυτό επειδή σήμερα ήδη οι πολίτες πρέπει, οι άνθρωποι πρέπει να μπορούν να αλλάξουν επάγγελμα και μάλιστα αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του βίου τους. Σας ευχαριστώ. Είναι και θέμα ταχείας έκφρασης. Μπορείτε κύριε υποψήφιε να γυρίσετε γιατί έχουμε την κυρία Κοράτσα Μπίλτ πίσω στη τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Εκτιμώ την αφοσίωση που δείξατε για την πρόθεση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και να σταματήσει ο κατακαιρματισμός. Υπάρχει κάτι κατεπήγον. Επεξεργαζόταν μια πράξη τρία της ενιαίας αγοράς. Ένα πλήρες πακέτο για να φύγουν οι διακρίσεις, οι περιορισμοί και τα εμπόδια και να υπάρχουν ισότιμες συνθήκες για το εμπόριο υπηρεσιών και αγαθών στην Ευρώπη Μπορείτε να παρουσιάσετε αυτό, αυτή την κίνηση το 2015. Δεύτερον, πάνω σε αυτά που είπε η Ρόζα Τούν όσον αφορά την περιαγωγή. Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο, ψηφίσαμε να μειωθεί το τέλος της περιαγωγής για τους πολίτες και όπως γνωρίζετε οι συνάδελφοί σας στο Συμβούλιο, οι πρώην Συμβουλοί σας τον μπλοκάρουν το όλο ζήτημα. Είσαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τη θέση σας του Αντιπροέδρου και πρώην Πρωθυπουργού για να έχετε σκληρή θέση και να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για τη μείωση των τελών περιαγωγής και να προωθεί το πακέτο για την ενιαία αγορά τηλεπικοινωνιών. Τρίτο ερώτημα που σχετίζεται. Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Είστε έτοιμο να αλλάξετε την οτροπία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να σκέφτεται ψηφιακά, δηλαδή να γνωρίσει ότι η καινοτομία ε, ε, είναι βοηθά στην πολιτική και καμιά φορά οι λιγότεροι κανόνες είναι καλύτεροι από υπερβολική ρύθμιση τόσο ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε και την ενιαία αγορά. Uh, λοιπόν, να δω τι σημειώσεις μου. Το τέλος περιαγωγής. Όλοι στην Ευρώπη περιμένουν την κατάργηση των υπερβολικών τελών περιαγωγής. Ήταν καλό για τον κόσμο όταν αυτά τα τέλη περιαγωγής μειώθηκαν για τα φωνητικά τηλεφωνήματα. Και γνωρίζω ότι πολλές από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών ήταν αρκετά ικανοποιημένες όταν συνέβη αυτό. Πριν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνουν αυτά τα μέτρα για την μείωση των τελών περιαγωγής. Οι περισσότερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών ήταν κατά αυτού. Είπαν ότι θα ήταν επιβλαβές. Τι συνέβη στην πραγματικότητα όμως. Ο κόσμος άρχισε να χρησιμοποιεί τα κινητά του τηλέφωνα και στο εξωτερικό, όταν πήγαινε διακοπές, στο εξωτερικό, όχι στην πατρίδα του. Και οι εταιρείε τηλεπικοινωνιών έχασαν όσον αφορά το περιθώριο κέρδους, αλλά κέρδισαν σε όγκο. Και ήταν υποφελές δεν λέω για όλες τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, αλλά για τις περισσότερες τηλεφωνικές εταιρείες. Τώρα, αναφερόμενοι στην κατάργηση των τελών περιαγωγής και για πληροφορίες, μετακίνηση πληροφοριών και στο διαδίκτυο, λένε για μία ακόμη φορά ότι αυτό θα είναι καταστροφικό για τις επιχειρήσεις. Το λένε κάποιες επιχειρήσεις, όχι όλες αλλά ελπίζω ότι ο κόσμος θα αρχίσει να χρησιμοποιεί πολύ περισσότερο τις κινητές του συσκευέ όταν ταξιδεύει στο εξωτερικό. Εγώ ίδιος ελέγχω αυτές τις δαπάνες, δεν πηγαίνω στις ίδιες ιστοσελίδες που επισκέφτομαι στην πατρίδα μου όταν είμαι εδώ. Πάρα πολύ γρήγορα πέρασε ο χρόνος και για να είμαι δίκαιο ο επόμενος από το SND ε, που θα θέσει την ερώτηση θα έχει περισσότερο χρόνο η κυρία Τόγια γιατί έδωσε περισσότερο λόγο, χρόνο στην κυρία Κορατσαμπέλ. Λοιπόν, θα ήθελα να σας αναφέρω ένα θέμα της ε, διακυβέρνησης στο διαδίκτυο. Η πολιτική μου ομάδα πέρα από το θέμα της ουτερότητας του δικτύου θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικότατο ρόλο και για τη διαφύληξη και σαν αντίβαρο όσον αφορά την διαχείριση του διαδικτύου κυρίως ε, από φορές φορεών που είναι εκτός της Επίρου που θέλουν να αφήσουν την επιλογή στους καταναλωτές. Ε, θέλετε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει πιο αποφασιστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή ο ρόλος Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι προθητικός για μια διακυβέρνηση του διαδικτύου που σέβεται την ελευθερία, τη δημοκρατία και εγγυάται την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Μετά το φάσμα το ραδιοφωνικό. Ε, ξεκίνησε να κάνει βήματα προόδου η ευρωπαϊκή πολιτική έχουμε, θέλουμε καλύτερη αποδοτικότερη χρήση του φάσματος αλλά για να αρμονιστεί το φάσμα και για να αποτελεσματική χρήση του θα πρέπει να θέσουμε το θέμα των αδειοδοτήσεων που τα κράτη-μέλη ε, το διαφυλάσσουν ως δική τους αρμοδιότητα. Και πιστεύουμε αντίθετα ότι πρέπει να είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ποια είναι η άποψή σας επί του θέματος, ευχαριστώ ευχαριστώ. Κάνοντας ε, λόγο για το εύρος συχνοτήτων και τον επιμερισμό, καταμερισμό αυτών, πολλά πρέπει να γίνουν. Όμως τα κράτη-μέλη γνωρίζουν ότι το εύρος αυτό, το φάσμα αυτό, είναι ένα είδος ε, φυσικού πόρου για αυτά. Και θέλουν αρκετά κράτη-μέλη να συλλέξουν το μέγιστο ποσό που μπορούν να συλλέξουν από τέτοιες ε, εισφορές. Ας κάνουμε λόγο τώρα για την τέταρτη γενεά ε, ηλεκτρονικών και ψηφιακών και να δούμε τι συμβαίνει. Σε κάποιες χώρες ε, LTE τέταρτης γενεάς καλύπτεται μεγάλο μέρος της επικράτειας από αυτού του είδους ε, της ε, ε, τεχνολογίας. Κάνω λόγος για τις χώρες της Σκανδιναβίας, σκανδιναβικές χώρες, σε σχέση με το 4G LTE. Σε άλλες χώρες είναι μηδενικό αυτό το ποσοστό. Δεν έχουν καν ξεκινήσει αυτές οι άλλες χώρες ούτε καν με τον επιμερισμό συχνοτήτων στο φάσμα, στο δίκτυό τους. Και αυτό πάλι βλέπουμε ότι αυξάνει τις διαφορές και τις ανισότητες μεταξύ κατών μελών. Και εδώ πρέπει να κάνουμε λόγο για συμφέροντα που υπάρχουν και που προστατεύονται από κάποιες χώρες. Σε κάποιες χώρες οι εταιρείε οι επικοινωνιών είναι τόσο ισχυρές και έχουν το πάνω χέρι που δεν έχουν κανένα συμφέρον να αλλάξει το πλαίσιο επενδύσεων που ισχύει και επικρατεί στις χώρες αυτές ε, σε σχέση για παράδειγμα με τις νέες τεχνολογίες. Σήμερα όμως ε, έχουμε ήδη την πέμπτη γενεά LTE ενώπιόν μας ε, ως προοπτική και όπως γνωρίζουμε αυτές οι προδιαγραφές αλλάζουν κάθε λίγα χρόνια. Μέγιστη λοιπόν ένα, μέγιστη εναρμόνιση, μέγιστος εναρμονισμός, κάνοντας λόγο για το φάσμα και τις συχνότητες. Είναι κάτι που χρειάζεται και χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερες δράσεις, αλλά και πολυπολική συνεργασία και όχι κατάχρηση εξουσίας. Ευχαριστώ. Thanks. We all know our country's best. Ναι, εμείς ξέρουμε τι καλύτερο για τις χώρες μας και τι είναι καλό για τις χώρες μας και λόγω του ίντερνετ τα πράγματα είναι αλήθεια ότι πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι λαμβάνοντας υπόψη αυτό που συμβαίνει στις χώρες μας κρίνουμε ότι αυτά τα πράγματα επεκτείνονται. Ο κόσμος όλο και περισσότερο χρησιμοποιεί το ίντερνετ και αυτό αφορά και τις επιχείρησεις και τους πολιτικούς. Αυτό που ήταν αδύνατο πριν από λίγα χρόνια είναι πραγματικότητα σήμερα και το σημαντικό σήμερα είναι βέβαια όχι μόνο να διασφαλίσουμε ότι θα είναι υπηρεσίε, αλλά το πώ θα έχουμε τι καλύτερε δυνατέ υπηρεσίε που θα αναπτυχθούν στον τομέα αυτό. Να σα ρωτήσω λοιπόν, ακολουθώντα με προηγούμενη, εισαγγίζουμε προηγούμενη ερώτηση, τι θα κάνετε ώστε να διασφαλίσετε ότι θα έχουμε το καλύτερο νομικό και τι ψηλότερε ταχύτητα στην Ευρώπη και το φάσμα που θα τα διασφαλίσει αυτό. Θεωρείτε ότι ο τωρινό στόχο επαρκεί ή θα πρέπει να πάμε παραπέρα. Ευχαριστώ. Uh, uh, Νομίζω ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί στην ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη είναι ήδη αρκετά φιλόδοξοι για να καλύψουμε, δηλαδή όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το 50%, 50 της Ένωσης μέχρι το 2020 με 100% εκατομμύρια να δευτερόλεπτο. Αυτό είναι αρκετά φιλόδοξο στόχος αλλά βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα 700 MHz για τα ψηφιακά δεδομένα. Αλλά όπως λέγαμε προηγουμένως, ξέραμε ότι αυτά τα 700 MHz που απαιτούνται για τα ευρωζωνικά δίκτυα, τα ψηφιακά, χρησιμοποιούνται διαφορετικά στις χώρες μέλη. Σε κάποιες χώρες μέλη χρησιμοποιούν αυτές τις συχνότητες για στρατιωτικούς σκοπούς. Για κάποιες λοιπόν χώρες οι γειτονές τους, μεγάλοι γειτονές τους, τους δημιουργούν προβλήματα. Γιατί αυτοί οι μεγάλοι γείτονε εκτός της Ένωσης χρησιμοποιούν αυτά τα 700 MHz για στρατιωτικούς σκοπούς και μεταδόσεις. Σε πολλές χώρες μέλη λοιπόν της Ένωσης τα 700 MHz χρησιμοποιούνται για τις μεταδόσεις. Οπότε και πάλι θα πρέπει να βρούμε συνενέσεις για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα 700 MHz με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Και βέβαια εκεί όπου ας πούμε τους μεταδότες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν άλλες συχνότητες πέρα αλλά των 700 και θα πρέπει να αποζημιωθούν. Αυτό είναι θέμα που αφορά τις χώρες μέλη αλλά ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πυγμή αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη εναρμόνιση και φιλόδοξους στόχους. Ευχαριστώ. Οι την Ήτρε Σοσιαλιστές πάλι. άκουσα προηγουμένως ότι μιλήσατε φιλανδικά, αλλά θα μιλήσω τώρα εγώ αγγλικά. Η νέα ψηφιακή αγορά παρέχει ευκαιρίες λοιπόν για οικονομική ανάπτυξη Χαίρομαι που τα αναφέρετε, αλλά βεβαίω υπάρχουν και κάποια τεχνολογικά ζητήματα. Τρει ώρε χρειαστήκαμε για να μιλήσουμε για την πέμπτη γενιά και εγώ θέλω να μιλήσω για το μέλλον. Όσο γίνεται ευρύτερη, ευρύτερα τα ευρυζωνικά, ευρυζωνικά δίκτυα για την ε, μετάδοση βίντεο και άλλων δεδομένων. Και ήταν από αυτούς που εθέτησαν την τρίτη γενιά πρώτη Ευρώπη, αλλά στην τέταρτη γενιά έμεινε πίσω. Για την πέμπτη γενιά θεωρείτε ότι είναι επιθυμά της δουλειά σα να προωθήσετε την υποδομή που θα αποτελέσει τη βάση για την ευρωπαϊκή κοινοτομία και ευκαιρίες και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις ώστε να διαναπτύσσουμε ηγετικό ρόλο και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας εδώ στην Ευρώπη. Thank I know that all the Finns... Ναι, ευχαριστώ. Και οι Εστονοί και οι Φιλανδοί και άλλοι είναι περήφανοι που η πρώτη γενιά δημιουργήθηκε το 1881. Η δεύτερη γενιά ήταν μια ιστορία επιτυχίας, success story για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάλι οι Φιλανδοί και οι Σουηδοί είχαν ηγετικό ρόλο. Τέταρτη γενιά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επαναλάβουμε και με την πέμπτη γενιά. Η Ευρώπη είχε πραγματικά ηγετική θέση παγκοσμίω. Αν τότε μπορούσαμε να το κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε και το 2020, όπου εμείς κατά πάσα πιθανότητα θα αρχίσουμε να χρησιμοποιήσουμε την πέμπτη, θα χρησιμοποιούμε την πέμπτη γενιά. Τώρα δεν έχουμε διακυβερνητικές ή διεθνείς συμφωνίες για την πέμπτη γενιά. Όμως οι επιστήμονες μας, οι μηχανικοί μας και οι πολιτικοί μας νομίζω ήδη προετοιμάζονται για την πέμπτη γενιά. Ελπίζω και αναμένω η πέμπτη γενιά να αφορά περισσότερο την αποτελεσματική χρήση. Δηλαδή το πώς θα χρησιμοποιούμε το φάσμα με ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο. Το πώς δηλαδή θα χρησιμοποιούμε την ενέργεια με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Δεν μιλάω εδώ για τις μπαταρίες και μόνο έτσι, αλλά η κατανάλωση ενέργειας το τομέα των τηλεπικοινωνιών και της κινητής τηλεφωνίας αυξάνεται. Οπότε αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα τώρα. Ευχαριστώ. Thank um, Τελευταίες πέντε ερωτήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε κυρία Σάντερ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, εδώ είμαι, εδώ είμαι οι γίγαντες του δικτύου ξεφεύγουν, α, λόγω διαφόρων περιπλόκων συστημάτων φορολογικών και κενών νομικών που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ξεφεύγουν λοιπόν γίγαντες. Η πρώτερη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολήθηκε με το θέμα ε, τοποθετώντα, δημιουργώντα μια ομάδα εμπειρογνωμόνων όσον αφορά τη φορολόγηση στο ψηφιακό τομέα και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σα όσον αφορά αυτό το θέμα θέτοντας τρία ερωτήματα. Πιστεύετε ότι είναι κανονικό να υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ των κερδών των ξένων ε, εταιριών και των πολύ χαμηλών φόρων που πληρώνουν. Δεύτερον, τι μέτρα θα θέλατε να λάβετε τόσο ώστε να αποφευχθεί το κοινωνικό dumping στο οποίο επιδίδονται τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως προς όφελος των επιχειρήσεων. Τρίτον, είσαστε υπέρ της φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών στα κράτη-μέλη στα οποία παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες. Ευχαριστώ. Thank ευχαριστώ. Μάλιστα. Η φορολόγηση είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα σήμερα. Κάποιες από τις πολυεθνικές μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν πολύ επιθετικού χαρακτήρα μορφές ε, φορολόγησης που επιλέγουν και που δεν είναι και πολύ θα έλεγα νόμιμες. Επιλέγουν τι μπορούν να κάνουν προς όφελός τους ε, στα διάφορα κράτη-μέλη και αυτό πράττουν. Και συνολικά χάνει έσοδα, υπάρχει απώλεια εσόδων στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. διαφυγώντα κέρδη, διαφυγώντας εισφορές λόγω φοροδιαφυγής. Να μην ε, υποτιμούμε λοιπόν ε, την ε, άποψη των πολιτών και την, α, τα δικά τους αισθήματα. Πρέπει να δημοσιοποιείται το πώς κάποιες εταιρείες φοροδιαφεύγουν και πώς αντιμετωπίζουν τα φορολογικά θέματα. Και δεν είμαι τόσο βέβαιος για το ότι οι φορολογούμενοι θα έχουν μια δική τους αντίδραση θετική. Θα είναι ιδιαίτερα αρνητική η στάση τους και η θέση τους για εκείνους που χρησιμοποιούν αυτές τις επιθετικές φορολογικές πολιτικές. Η φοροδιαφυγή και πάλι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα τεραστίων διαστάσεων πρόβλημα. Και πάλι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, αυτά τα θέματα. Και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Αποκινούμε τον Επίτροπο κύριο Πιέρ Μοσκοβισή ώστε να αποφύγουμε τέτοιου είδους ε, φαινόμενα φοροδιαφυγής, να αποφευθεί η φοροδιαφυγή. Και είμαι υπέρ και της, ε, του ενιοποιημένου ε, εταιρικού φόρου που θα ισχύει στην Ευρώπη. Αυτή η πρόσθετη εναλλακτική δυνατότητα θα δημιουργήσει πρόσθετες δυνατότητες ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να δρουν σε ένα έντιμο πλαίσιο και να είναι έντιμες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έξοχη προφορά του ονόματο την προηγούμενη φορά καλύτερα από πολλούς άλλους. Υποψήφιε επίτροπε, προστασία δεδομένων, ίσως για τελευταία φορά σε αυτή την ακρόαση να το θίξουμε. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Μία γενική και μία ειδική. Γενική. Λοιπόν, το ψηφιακό θεματολόγιο είναι πάρα πολύ ευρύ. Πώς θεωρείτε ότι είναι δυνατόν να καλυφθούν όλα αυτά, πώς θα διοργανώσετε ένα νομικό πλαίσιο ούτω ώστε προστασία των δεδομένων και προστασία τη ιδιωτική ζωή πάντα να θεωρούνται ότι έχουν ύψιστη προτεραιότητα σε όλο το θεματολόγιο. Δεύτερον, άκουσα προσεκτικά Η είπατε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ εμπορικών συμφερόντων και προστασία δεδομένων. Εγώ δεν βλέπω αυτή την ισορροπία. Η προστασία των δεδομένων είναι το ουσιαστικό κομμάτι του ζητήματος. Πάντα πρέπει να υπάρχει ισορροπία, αυτό πιστεύετε και εσείς όσον αφορά την προστασία των δεδομένων έχετε κάποιες, κάποια όρια, κάποιοι κόκκινες γραμμές όπου λέτε τέρμα ισορροπία, μετράει η προστασία των δεδομένων και τίποτα άλλο. Έχετε αυτές τις ερυθρές γραμμές, αυτές τις διαχωριστικές και ποιε είναι αυτές. Απάντηση, η προστασία των δεδομένων είναι απόλυτη αξία. Είναι η βάση για όλες τις ψηφιακέ λύσεις. Αν δεν προστατεύονται σωστά τα δεδομένα με ασφάλεια, καμία επιχείρηση δεν θα χρησιμοποιεί, δεν θα χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, τις υπηρεσίες. Είναι προαπαιτούμενο. Η προστασία των δεδομένων πρέπει να παραμείνει ύψιστη προτεραιότητα. Δεν νομίζω και λυπάμαι που το λέω, πρέπει να διορθώσω αυτά που είπα. Πρέπει να βρει κανείς κάποια ισορροπία μεταξύ εμπορικών συμφερόντων και προστασία των δεδομένων. Διορθώ τον εαυτό μου. Για να βρει όμως... Για να βρει κανείς την ισορροπία μεταξύ συμφερόντων εμπορικών και προστασία δεδομένων είναι κάτι απαραίτητο. Και για την υγεία, το αναφέραμε πριν στην, όσον αφορά ε, την έρευνα να θεσπίσουμε κάποιους κανόνες που θα μας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε τη σωστή προσέγγιση για την έρευνα. Σε κάποιες χώρες, στις ΗΠΑ, παραδείγματος χάρη, είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει κανείς Ανείχνευση γίνεται στην Ιαπωνία. Uh, uh, Για να γίνεται ανείχνευση στοιχείων, εξόριξη στοιχείων ηλεκτρονικά. Αυτό γίνεται σε άλλες χώρες, αλλά όχι στην Ευρώπη. Πρέπει να βρούμε λύσεις που να επιτρέπουν στα ερευνητικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια να ασχοληθούν με το θέμα αυτό της προσπάθειας εξερεύνησης στοιχείων, άντλησης στοιχείων και πληροφοριών. Το ΕΛΚ τώρα έχει το λόγο. Ο κ. Μπόνι. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, η οριζόντια προσέγγιση είναι κλειδί για μια ψηφιακή στατηγική. Χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων και των πτυχών Τη ενιαίας αγορά. Έχουμε την προστασία των δεδομένων, θέλουμε ανάπτυξη δεδομένων, ανοιχτή προσβασιμότητα στα στοιχεία και ασφάλεια των δεδομένων. Όλα αυτά μαζί πρέπει να κινηθούν. Χρειάζεται ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων των πολιτών για την προστασία της ιδιωτική ζωής, τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Πρέπει να εφαρμοστούν όλα μαζί. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων αλλά δεν χρειάζονται υπερβολικά άχθη. Χρειάζεται καλύτερο κλίμα για, την, για το άνοιγμα των στοιχείων και τη διάδοσή τους. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή ενημέρωση και χωρίς πληρωμές διατίθεται οι πληροφορίες ελεύθερα στους πολίτες. Χρειάζεται ελευθερία και ασφάλεια στα δίκτυα, να ανταποκρινόμαστε στις κυβερνοαπειλές και χρειαζόμαστε κοινά ευρωπαϊκά εργαλεία. Πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε σωστά συντονισμένη πολιτική για να εφαρμοστεί νέα ψηφιακή στρατηγική και πώς θα πείσετε τα κράτη-μέλη να είναι πιο ανοιχτά για εναρμόνιση των νομοθεσιών σε βασικούς τομείς της ψηφιακής ενίας αγοράς και να υπάρχουν δεσμευτικές λύσεις, κυρίως όσον αφορά την προστασία, την ασφάλεια και τη διαβίβαση και το μοίρασμα των στοιχείων. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Συζητήσαμε σήμερα επανειλημμένα πολλές φορές ήδη για τα θέματα ασφάλειας της προστασίας δεδομένων και δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα ήδη προανέφερα προηγούμενα. Αναφέρατε τα ανοιχτού χαρακτήρα δεδομένα, open data. Πιστεύω ότι όλα αυτού του χαρακτήρα στοιχεία που συλλέγονται για την παραγωγή εσόδων από πλευράς χωρών μας πρέπει να είναι ανοιχτού χαρακτήρα για την εμπορική χρήση ή μη. Είναι δυνατόν λοιπόν να βρούμε αντιστοιχίες, αντιστοίχηση χρησιμοποιώντας τέτοιου είδους ανοιχτά χρη, ε, χρηστικά στοιχεία που θα είναι επωφελή για την κοινωνία μας, για τους πολίτες μας και αυτή η πρωτοβουλία θα είναι υποφελής. Ο κόσμος γίνεται όλο και περισσότερο ηλεκτρονικός και κινείται από τα δεδομένα και τρέφεται από αυτά τα δεδομένα. Οι επιχειρήσεις μας τρέφονται και ζουν, επιβιώνουν μέσω αυτών των στοιχείων. Πάνω ένα τεράστιο ποσοστό της παραγωγής βασίζεται σε αυτά τα ψηφιακά οι αυτοκινητοβιομηχανίες ήδη μπορούμε να πούμε σήμερα ότι οι αυτοκινητοβιομηχανίες μας είναι ψηφιακές βιομηχανίες ήδη σήμερα. Ας πάρουμε την φαρμακοβιομηχανία. Δεν είναι πια χημικής, ε, χημικού χαρακτήρα βιομηχανίες. Είναι επιχειρήσεις και βιομηχανίες ψηφιακές ήδη σήμερα. Μπορεί κανείς να προβλέψει πως ε, ο μοριακός χαρακτήρας συγκεκριμένων στοιχείων μπορεί να συνδυαστεί χωρίς χημικούς τύπους ή χωρίς χημεία, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά δεδομένα, ψηφιακά δεδομένα και τέτοιου είδους data, στοιχεία και δεδομένα. Η προστασία και πάλι των δεδομένων, data protection, έχει θεμελιώδη σημασία για όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουν τέτοια σπουδαιότητα για τις βιομηχανίες, επιχειρήσεις και την κοινωνία μας. Ευχαριστώ. Από την Επιτροπή Πολιτισμού. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα μιλήσω ιταλικά. Κύριε Αντσίπα. Ω τη Επιτροπή Πολιτισμού, ρωτώ κατά την εφαρμογή της ενιαίας ψηφιακής αγοράς στην Ευρώπη θα δεσμευθείτε να προωθήσετε την ιδιαιτερότητα των πολιτιστικών περιεχομένων και την προώθηση τηλεοπτικών προϊόντων στο ίντερνετ ως επίσης και σημαντικό πόρο για την αξιοποίηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και την ασφάλιση ανάπτυξη και θέσεων Για μας αυτό σημαίνει ότι Πρέπει να υπάρξει μια οδηγία που θα προστατεύει όμως την επέκταση αυτών των μορφών επικοινωνίας στο ίντερνετ. Και θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζει και την σωστή αμοιβή των δημιουργών. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε ποιες δεσμεύσεις θα αναλάβετε. Τέλος, μας είπατε κάποια πράγματα για την ηλεκτρονική φορολογική διακυβέρνηση όμως να μας πείτε τι γίνεται και για το τι θα πρέπει να γίνει για να αποφευχθούν δεσπόζουσε θέσει και στο τομέα του πολιτιστικού περιεχομένου, όπου ακριβώ δεν γίνονται επενδύσει ευρωπαϊκέ, χρησιμοποιούνται αυθαίρετα πνευματικά δικαιώματα και υπάρχει παρασυντική κατάσταση σε σχέση με την πολιτιστική παραγωγή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη που παραβαίνουμε τους κανόνες, αλλά ήταν ε, σημαντικό να ακούσουμε και την Επιτροπή Πολιτισμού. Σας άφησα παραπάνω, αλλά ήταν χρήσιμο. Σας ευχαριστώ, λέει η κυρία Κώστα. Ναι, η πολιτιστική πολυμορφία στην Ένωση είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι και θα πρέπει να την προστατεύσουμε αυτή την πολιτιστική πολυμορφία της Ένωσης ο τομέας των οπτικοακουστικών και του πολιτισμού δημιουργεί το 4% του ΑΕΠ της Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό τμήμα αυτό. Έστω και αν μιλούσαμε καθαρά για οικονομικά στοιχεία. Η βασική λοιπόν αξία όμως, εδώ, η υποκειμένη είναι η, ο πολιτισμός ο ίδιος. Για τις υπηρεσίες over the top αυτές δεν ακολουθούν κανονισμούς για τα πνευματικαιώματα ας πούμε. Και μάλιστα δεν μπορούν να το πράξουν επειδή η δομή αυτών των υπηρεσιών over the top δεν μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία. Υπάρχει βεβαίως ένα είδος ανισοκατανομής μεταξύ υπηρεσιών over the top και οργανισμών τηλεπικοινωνιών. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα σωστό πρότυπο, ένα σωστό μοντέλο. Το πώς θα μπορούσε να υπάρχει καρποφόρα διάδραση μεταξύ των δύο. Σήμερα οι, οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών είναι υπεύθυνοι ας πούμε για τις ευρωζωνικές ε, υπηρεσίες. Όμως οι over the top υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις υπηρεσίες, όμως δεν είναι υπεύθυνε για δημιουργήσεις αυτών των δικτύων αλλά και πάλι παραχωμένοι στο θέμα του πολιτισμού. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε το δημιουργικό μας τομέα, θα πρέπει να υποστηρίξουμε την παραγωγή ταινιών, την κινηματογραφία, γιατί ακριβώς θα πρέπει να προσπίσουμε την ε, πολιτιστική πολυμορφία της Ένωσης. Ευχαριστώ. Τελευταίο αλλά έσχατος, από την Επιτροπή Πολιτισμού. Τελευταία ερώτηση. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, κάνετε λόγο για μια δυναμική παρέμβαση για την ψηφιακή αγορά. Πώς αξιολογείτε τον ρόλο του δημιουργικού, παραγωγικού, καλλιτεχνικού τομέα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τον διτό χαρακτήρα του πολιτισμικού προϊόντος οικονομικού χαρακτήρα και κοινωνικού χαρακτήρα προϊόντος. Πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ των οικονομικών χαρακτηριστικών και των κοινωνικών χαρακτηριστικών και πώς συγκεκριμένα θα αντιμετωπίσετε τις αυξημένες προκλήσεις σε σχέση με την ψηφιακή αγορά και τις διαφορετικές δυνατότητες ρύθμισης που υπάρχουν. Πώς αντιμετωπίζετε την γεωγραφική κατάτμιση, τον, τον κατακαιρματισμό ε, γεωγραφικά και πώς θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε αυτή αυτή την κατάσταση. Thank Σας ευχαριστώ. Ο πολιτισμός, τα πολιτισμικά προϊόντα και τα ψηφιακά προϊόντα δεν είναι εχθροί, είναι σύμμαχοι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολλά καλά θετικά παραδείγματα όπου αυτή η συνεργασία μεταξύ πολιτισμού και ψηφιακών είναι πολύ καρποφόρα, γόνιμη. Για να το δούμε αυτό. Έχουμε μια ιστοσελίδα για παράδειγμα που μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση από όλα τα κράτη-μέλη σε αυτήν και μπορεί να χαρεί τον, την πλούσια πολιτισμική κληρονομιά μας. Πάνω από 30 εκατομμύρια αντικείμενα υπάρχουν σε αυτή τη συλλογή, στην Ευρωπαϊάνα, σε αυτή την ιστοπύλη και τα ψηφιακά παρέχουν μέσω της Ευρωπαϊάνα πολλές δυνατότητες για την προαγωγή των πολιτισμικών και πολιτιστικών μέσω των ψηφιακών βιβλιοθηκών για παράδειγμα, ψηφιακών μουσείων και ψηφιακές ε, δυνατότητες ε, και διευκολύνσεις για την προαγωγή του πολιτισμού μας. Ψηφιακά μέσα για την προστασία επίσης ε, της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Και όπως προανέφερα στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις, είμαι κατά της γεωγραφικής, ας το πούμε έτσι, εμ, ιδιαιτερότητας θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τις διατάξεις μας για τα ψηφιακά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα της εδαφικότητας. Είναι πολλά από αυτά ανεδαφικά και πρέπει να επικαιροποιηθούν. Ωστόσο, θα ολοκληρώσω με μια παρατήρηση ως εξής. Ως φορολογούμενος πλήρωνα για τα ποδοσφαιρικά, τις ποδοσφαιρικές συναντήσεις και τους αγώνες ποδοσφαίρου στην Εστονία. Εδώ όμως στο Βέλγιο δεν είχα πρόσβαση σε αυτού του είδους τα παιχνίδια. Γιατί ούτε καν είχα πρόσβαση τα κύρια προγράμματα ε, δελτίων ειδήσεων διότι είχαν τροχοπεδηθεί, είχαν, υπήρχαν προβλήματα και δεν μπορούσαν να αναμεταδοθούν αυτά τα δελτία ειδήσεων. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι σωστό και δίκαιο δεν μπορούμε να δεχθούμε ένα τέτοιο, ε, χαρακτήρα γεωγραφικής ε, διακριτικής αρνητικής μεταχείρισης, ας το αποκαλέσω έτσι. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον υποψήφιο επίτροπο για όλες τις απαντήσεις του και σε ευχαριστώ για τις πολλές, ποικίλε και ποικιλόμορφες ερωτήσεις που προήλθαν από τα μέλη τεσσάρων πιτροπών απόψε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, έχετε τώρα την ευκαιρία για ένα πεντάλεπτο να συνοψίσετε και θα σας πω τι θα γίνει στη συνέχεια. Έχετε πέντε λεπτά για τελικές δηλώσεις.